Przepraszam za opóźnienie, ale no tak się złożyło trzy komisje. Αγαπητοί συνάδελφοι, τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, συνεταιρίασαν για να μιλήσουν για ένα σημαντικό θέμα. πάρα bardzo ευχαριστώ. Ας δώσταμε ρουμένιτσου rumieńców z tego tytułu. Σας ευχαριστώ. Μπαίνουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, στην παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, Αγκρή, για την κρίση των δημητριακών και άλλων καλλιεργειών Δεν ξεχνάμε τη συζήτηση που κάναμε για τον γαλακτοκομικό τομέα, των ποροκυπευτικών, του χείριου κρέατος, τα διάφορα προβλήματα των διαφόρων τομέων και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα άλλο σημαντικό θέμα που αφορούσε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, που έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και μιλάω πιο συγκεκριμένα για τα προβλήματα των Δημητριακών. Η Γαλλία, η Γερμανία επλήγησαν οι εισοδιές μειώνονται. Υπάρχει και μια μείωση της ποιότητας των δημητριακών και αυτό έχει επίπτωση στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς δημητριακών, εξού και το αίτημα που μας υποβλήθηκε. Μάλιστα ήταν αίτημα της κυρίας Μαγκίνες. Την υποστήριξαν και οι συντονιστές. Να εγγύψουμε περισσότερο στην κατάσταση της αγοράς των δημητριακών. Θα δώσουμε το λόγο λοιπόν τώρα στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, στον Γενικό Διευθυντή, στον Διευθυντή, συγγνώμη, ο οποίος είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό και ο οποίος θα μας παρουσιάσει την κατάσταση όπως έχει σήμερα στην αγορά. Κύριε Διευθυντά, σας δίνω το λόγο. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή που έβαλε αυτό το σημαντικό θέμα στη μερίσια διάταξη. Και εμεί το εξετάζουμε πολύ προσεκτικά στη Γενική Διεύθυνση Γεωργία. και χαίρομαι που ήρθα εδώ για να σα εξηγήσω σύντομα πώ βλέπουμε εμεί την κατάσταση. Πρέπει να ξεκινήσω με μια διαπίστωση, αν κονστά όπω λέμε στα γαλλικά, ότι τα δημητριακά εισοδιά του 2016 ήταν πολύ χαμηλότερη από τι προσδοκίε μα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει και ποσοτικά, τον όγκο δηλαδή της παραγωγής, αλλά και για την ποιότητά της. Να σας δώσω ένα νούμερο. Οι εκτιμήσεις μας σήμερα είναι ότι η σοδιά θα είναι περίπου 294 εκατομμύρια τόνοι, που είναι 5% λιγότερο από ό,τι το 2015 και 3% λιγότερο από το μέσο όρο της πενταετίας. Με αυτά τα νούμερα θέλω να κάνω δύο άλλες παρατηρήσεις. Ε, για μία μεικτή εικόνα. Αυτά τα νούμερα είναι πανευρωπαϊκά νούμερα. Όταν πηγαίνουμε τώρα στις ε, σοδιές και στα κράτη-μέλη, στις διάφορες περιφέρειες, η επίπτωση, η κατάσταση διαφέρει πολύ περισσότερο. Γιατί έτσι ας δούμε όρους. Η Γαλλία, ας πούμε, ε, πλήγει περισσότερο. Και αυτό έχει ουσιαστική επίπτωση στα νούμερα, γιατί όπως ξέρετε η Γαλλία είναι ο βασικός παραγωγός σιτηρών και μαλακού σίτου στα κράτη-μέλη. Και αυτό οφείλεται λόγω των άσχημων κλιματικών συνθήκων και σε πολλές ασθένειες στο τέλος της περίοδου ανθοφορίας. Λόγω κακού καιρού λοιπόν και λόγω ασθενειών, είχαμε τη χαμηλότερη απόδοση στη Γαλλία τα τελευταία 30 χρόνια. Φέτος, το 16 δηλαδή. Μείον 24% το 2016 σε σχέση με το 2015. Τη συνολική παραγωγή των σιτηρών μιλάω. Τώρα, ο μαλακός σίτος, για να δούμε ειδικά το μαλακό σίτο, είναι ακόμα περισσότερο. Είναι 31% λιγότερο από ό,τι πέρυσι το 2015, στη Γαλλία αυτό, έτσι. Άλλα κράτη-μέλη τώρα. Και αυτά είναι σε αντίστοιχη κατάσταση. Θα ήθελα να αναφέρω εδώ τη Δανία, την Εστονία, την Κύπρο, τη Λετωνία. Πάνω κάτω 20% λιγότερο σε σχέση με τη σοδιά του 2015, είχαμε φέτος, αλλά και το Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και τη Λιθουανία. Αν κοιτάξουμε τις διάφορες οδιέ, τις διάφορες καλλιέργειες. Ε, ο ΣΥΤΟΣ ε, επηρεάστηκε από χαμηλές αποδόσεις κυρίω μείον 11% σε σχέση με το 2015, ενώ ε, το κρυθάρι είναι μείον 4% και το, ο αραβόσιτος αυξήθηκε σε σχέση με το 2015, συν 8%. Ο μαλακός είναι η πιο σημαντική εισοδιά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου το 50% των σιτηρών συνολικά. Είναι ο μαλακός σύτος, ο σύτος, περιπτώσει. Εξού και αυτή η δραματική κατάσταση με τα νούμερα. Ε, ο ραβόσιτος και, στο, και το κρυθάρι δεν είναι τόσο προβληματικά σιτηρά. Α, αυτή η κακή κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη ε, έρχεται σε αντίθεση από σχετικά καλές αποδόσεις σε άλλα κράτη-μέλη όμως, κυρίως. Στην νότια και Ανατολική Ευρώπη. Με βάση τις τελευταίες προβλέψεις η εισοδία ήταν καλή, για να μην πω και φανταστική. Με τρομερές σωθίες μερικές φορές ε, σωθίες. Ισπανία, Ουγγαρία, Σλοβακία. Το 2016 στα σιτηρά θα, είχα, θα έχουμε 20 με 25% παραπάνω απόδοση από ό,τι το 2015. Και αυτό εξηγεί ότι αν κοιτάξετε τη συνολική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι προφανώς αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική που καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι η εισοδιά είναι μόνο κατά τη κάτω τα 300 εκατομμύρια τόνους ε, του μέσου όρου της πενταετίας. 3% δηλαδή ε, λιγότερο από το μέσο όρο της πενταετίας και 5% παρακάτω από το 2015. Αυτό το νούμερο με, το με τα υψηλά αποθέματα στις αρχές της ε, περίοδου εμπορίας ε, τελικά μπορούμε να πούμε ότι εξορροπείται η αγορά και μπορεί να ανεφοδιαστεί από τις αποθήκες που έχουμε. Η άλλη απόφαση που θέλω να βάλω στη συζήτηση, Πρόεδρε, είναι ότι η εισοδιά του 2016 ήταν πολύ πτωχή. Είχαμε τρία καλά χρόνια πριν, με τρομερές παραγωγές, υψηλότατες, πάνω από τους 300.000 ε, ε, τόνους το 13, 14 και 15 είχαμε τέλειες αποδόσεις. Όταν δούμε τις ε, τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να σας πω ότι η αγορά των σιτηρών είναι μια παγκόσμια αγορά. Οι τιμές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις τιμές παγκόσμιας αγοράς. Είναι μια παγκόσμια λοιπόν αγορά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τη ροή της παγκόσμια αγορά. Και ενώ είμαστε σημαντική παραγωγή, δεν είμαστε οι μόνοι οι οποίοι καθορίζουμε την κατάσταση των σιτηρών στον πλανήτη. Παρότι λοιπόν οι τιμές έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια παγκόσμια, παρόλα αυτά είναι αρκετά ψηλότερα από τις τιμές της παρέμβασης. Δηλαδή είναι πάνω από 50% υψηλότερε από τι τιμέ τη παρέμβαση. Και αυτό είναι σημαντικό, νομίζω, γιατί είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση στα σιτηρά από ότι ας πούμε το γαλακτοκομικό τομέα ή τα ζώα, τα τυγνοτροφία δηλαδή, όπου θα θυμάστε, θα θυμάστε ότι το σύστημα παρέμβασης έχει χρησιμοποιηθεί. Ε, τα προγράμματα παρέμβασης στα σιτηρά δεν έχουν ε, χρησιμοποιηθεί από το, 12, από το 2010 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η παραγωγή μας, οι έμποροι μας είναι πολύ ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια χώρα. Και αυτό φαίνεται και από τις ε, καταπληκτικές ε, εξαγωγές των σιτηρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2014 και το 2015 οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ πάνω από 50 εκατομμύρια τόνους. Και πέρυσι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο πρώτος εξαγωγέας παγκόσμια και για το κρυθάρι και για το ΣΥΤΟ. Αν δείτε την αξία αυτών των εξαγωγών, ε, στο ΣΥΤΟ φτάσαμε στα 6,34 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι παν 5% περίπου των συνολικών εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το τρίτο ε, γεωργικό προϊόν που εξάγεται μετά τα κρασιά και τα αλκοολούχα. Εάν μειωθούν οι τιμές στην παγκόσμια αγορά, ε, που, αυτό που βλέπουμε σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, η επίπτωση θα γίνει αισθητή πάρα αυτά και εσωτερικά, γιατί δεν υπάρχει πια διαφορά. Με τις τιμές ε, αυτή τη στιγμή περίπου στα 150 με 160 ευρώ ανατόνο, έτσι, 150 με 160 ευρώ ανατόνο για το μαλακό σίτο, ε, υπάρχει ένα πρόβλημα για τους Ευρωπαίους καλλιεργητές. Συνοψίζοντας, Πρόεδρε, τι μπορώ να πω. Ότι ενώ οι τιμές έχουν να μειωθεί παγκόσμια και επομένως και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Παρ' όλα αυτά, πολύ πάνω από τις τιμές παρέμβαση ακόμα. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε και κάποιους ε, παράγοντες ε, που αλλάζουν την, την εικόνα. Παραδείγματο χάρη, ε, το κόστος παραγωγής για τους γεωργούς έχει μειωθεί σημαντικά. Ειδικά όταν κοιτάμε τις τιμές των λοιπασμάτων, που είναι σημαντικό έξοδο για τους γεωργούς, είναι σημαντικό τμήμα του, των εξόδων τους. Έχουν μειωθεί κατά 50% τα τελευταία δύο χρόνια οι τιμές αυτές των λοιπασμάτων κτλ. Λογική συνέπεια, ας πούμε, των χαμηλότερων τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου και επομένως βοήθησαν για να διατηρήσουν ας πούμε, τα περιθώρια κέρδους των διοργών. Να υπενθυμίσω επίσης ότι υπάρχουν προγράμματα στο εσωτερικό της κοινή γεωργικής πολιτικής που προβλέπουν σημαντική υποστήριξη ε, σε, με πληρωμές που βασίζονται στις επιφάνειες, ε, στήριξη του δεύτερου πυλώνα και αν κοιτάξουμε τις ε, μέσα στη μέση Ευρωπαϊκή Ένωσης. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, αλλά οι άμεσες πληρωμές ε, κατά μέσο όρο για τις αρωτρές καλλιέργειες είναι περίπου 260 ευρώ ανά εκτάριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, πέρα από αυτήν την ενίσχυση, τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να ξεκινήσουν τα δικά τους μέτρα ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, στα πλαίσια βέβαια των κανόνων και με σεβασμό των κανόνων κρατικών ισχύσεων. Και για να βοηθήσουν τους γεωργού ε, Δημητριακών, η Γαλλία ξεκίνησε ένα σύστημα δημοσίων εγγύσεων για να τους βοηθήσει να επιβιώσουν αυτή την ε, δραματική πτώση των ε, εισοδημάτων τους και να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος σε καλύτερα επιτόκια από αυτά που προσφέρουν οι τράπεζες, ας πούμε. Ε, κοιτάμε αυτό το πακέτο της Γαλλίας αυτή τη στιγμή. Επομένως, συμπερασματικά, παρά την κακή χρονιά, αναμφίβολα, για τους γεωργούς σιτηρών και μια αυξημένη αστάθεια, πιστεύουμε ότι ο τομέας των σιτηρών είναι σε σχετικά καλή κατάσταση ακόμα. Φυσικά, αν το συγκρίνουμε με άλλους τομείς, και υπάρχει μια μεγάλη διαφορά εδώ, είναι ότι ενώ η αστάθεια στις αγορές προφανώς υπάρχει για τα σιτηρά, ε, ο τομέας των σιτηρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει διαφορετικά ελλείμματα, προβλήματα. Δεν πλήττεται από τα διαφορετικά μακροχρόνια προβλήματα που ταλανίζουν άλλους τομείς που συζητάμε συχνά εδώ. Η παραγωγή μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, έχουν ένα καλό ανεπτυγμένο τομέα και διαχειρίζονται καλά τους κινδύνους τους. Ε, τα future ε, τα χρησιμοποιούν σε πολύ ευρία κλίμακα, ας πούμε, για τα σιτηρά τα παράγωγα future. Και επίσης έχουν και άλλες διατάξεις ε, στα πλαίσια της ε, ΚΟΑ, της κοινή οργάνωσης αγοράς. Επομένως, για τα σιτηρά ε, είμαι αισιόδοξο, θα πρέπει να, είμαστε, έχουμε το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, αλλά όπως είπε και η Διευθυντική Κομισιόν, θα πρέπει να μάθουμε από αυτές τις κρίσεις, από αυτές τις κακές χρονιές και να σκεφτούμε πώς η μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020 μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα για να ενισχύσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γεωργίας. Με καλύτερη διαχείριση του κινδύνου κυρίως. Αυτά τα θέματα τα σκεφτόμαστε και θα επανέλθουμε σε αυτά και θα θέλαμε να τα συζητήσουμε μαζί σας. Φυσικά θα πρέπει να αναφέρω ότι στο δεύτερο πυλώνα της ε, ΚΑΠ υπό τον κανόνα για την ανάπτυξη της ε, υπαίθρου υπάρχει ένα ταμείο για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων που είναι στη διάθεση των κρατών μελών και ο Επίτροπος, μάλλον η Κομισιόν καλύτερα, ως τμήμα της πρότασης για το γενικό κανονισμό του Omnibus έκανε μια πρόταση για να εισαγάγει περαιτέρω ευελιξία στα κράτη-μέλη ώστε να μπορούν πιο εύκολα να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο για τους γεωργούς. Και είμαι σίγουρο ότι η Κομισιόν ε, θα σας πει περισσότερα σε λίγο για αυτό το θέμα του Omnibus. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να σας εξηγήσω την άποψή μας για την αγορά των σιτηρών που δεν είναι και τόσο καλή και την οποία παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον και, και εκ του συνεγγύς. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Οκτώ συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ένα μισή λεπτό καθένας παρακαλώ. Γιατί στι ε, πέντε θα έρθει και ο Επίτροπο. Ένα μισή λεπτό λοιπόν ο καθένα. Η κυρία Μαγκίνε πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για την παρουσίαση αυτή και που μα έβαλε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη τόσο σύντομα. Να ευχαριστήσουμε και του συντονιστέ. Είναι σημαντικό το γεγονό ότι οι αγρότε μα ακούν τώρα να μιλάμε για τα θέματα που του απασχολούν τώρα, όχι σε ένα χρόνο. Και χαίρομαι ότι αναγνωρίζουμε για το ότι αναγνωρίζουμε ότι είναι κακή η χρονιά αυτή. Από τα ταξίδια μου στην Ιρλανδία να σα πω ότι ήταν φρικτή η σουδιά. Και φυσικά αυτό έχει και ψυχολογικέ επιπτώσει. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει και με τη διαχείριση του κινδύνου. Αυτό μας λένε λοιπόν πλέον οι αγρότες. Τι μπορεί να γίνει από πλευρά πολιτικής για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση του κινδύνου σε ό,τι αφορά την αντικτύπωση στην αγορά και την ε, στρέβλωση που προκαλείται στην αγορά. Κατά δεύτερο, δεν αναφέρθηκε κατά πόσο α, υπάρχει ενίσχυση άμεση των αγροτών και προφανώς θα πρέπει να αντιποκρίνεται η Ευρώπη στις ανάγκες ε, των γεωργών. Αν λοιπόν η αγορά των σιτηρών είναι παγκοσμιοποιημένη, χρειάζεται να ξέρουν ότι αυτή η... αυτός ο χαρακτήρας διακυμάνσεων και βαλωτότητας μπορεί να γίνεται να είναι διαχειρίσιμος σε παγκόσμιο επίπεδο και θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσει να επιτευχθεί αυτό καλύτερα στο μέλλον. Για την αντιμετώπιση της αστάθειας δηλαδή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονό ότι δείχνει τόσο μεγάλη κατανόηση μία βουλευτή ε, τη ε, Ιρλανδία για τα προβλήματα τη Γαλλία. Ο κ. Ραπέ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πλήττει πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και οι χώρες της Βαλτικής. Έχουμε και το... Και έχουμε και τη μονάδα των η οποία επίση επιδεινώνει την κατάσταση. Άρα λοιπόν ε, πρέπει να σα πω ότι έχουν πληχθεί όλοι οι τομεί, μεταξύ των οποίων και ο τομέα των δημητριακών που χρησιμοποιούνται και για ζωοτροφές. Έχουν μειωθεί τα εισοδήματα έως και δύο φορές σε σχέση με το περσινό έτος. Και ο κόσμος φυσικά έρχεται και ρωτάει τι μπορεί να γίνει. Γιατί δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα ευρωπαϊκά έργα, δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνειά τους, δεν μπορούν να ανταποκριθούν και στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει δεν έχουν και δυνατότητα να το ρυθμίσουν από πλευρά των προμηθευτών. Κάτι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε εδώ και τώρα, σήμερα, όχι το 2020 και μετά, όπως μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι να το κάνουμε το 2020, τώρα πρέπει να βρούμε λύσεις. Γιατί όταν λέμε ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πέσει κατά ε, λίγες ποσοστιαίες μονάδες. Ε, αυτό δεν μας αρκεί. Δεν ε, αρκεί αυτό για τις χώρες μας που έχουν πληχθεί πιο πολύ από κάθε άλλη. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω και θα πρέπει να αποσταλεί ένα μήνυμα προς τα κρατημέλη από πλευρά της Επιτροπής για να χρησιμοποιηθούν να επιπρόσθετα μέτρα και να βοηθηθούν άμεσα οι αγρότες. Ο κ. Φλάνεγκαν. Ευχαριστώ. Και αυτό που ακούω και αυτό που αντυχεί στα αυτιά μου είναι ότι δεν θα δοθεί άμεση βοήθεια. Αυτό ψάχνει ο κόσμος, αυτό ψάχνουν οι αγρότες στην Ευρώπη. Εντάξει, ωραία, το βάλαμε στην ατζέντα, πολύ ωραία, αλλά πώς θα βοηθήσει αυτό τους αγρότες. Το ότι καθόμαστε και το συζητάμε, δηλαδή εμείς δημόσια, πώς θα βοηθήσει. το, τον κύκλο. Αυτό προσπαθείτε να κάνετε. Μα λέτε ότι η παραγωγή είναι σε μια ανταγωνιστική αγορά, λοιπόν. Αυτό από ό,τι φαίνεται το αντιμετωπίζουμε θεωρητικά. Στην πράξη το αντιμετωπίζουμε. Όχι. Γιατί αυτή η ιδέα ότι αν υπάρχει κάποια επιπλέον περιθώρια το α, ωφελείται ο αγρότης, αυτό είναι πραγματικά ανοησία. Γιατί έγινε τίποτα τέτοιο όταν έπεσαν οι τιμές των λοιπασμάτων. Εξηγήστε μας λοιπόν πώς είναι βιώσιμο το γενικό αυτό. Όταν ένας αγρότης 19 χρονών βλέπει να χάνετε όλη του εισοδιά, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μπορεί να μας πει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί να παίζουν ρώσικη ρουλέτα οι αγρότες. Δηλαδή όταν κερδίζουν χάνουν και όταν χάνουν καταστρέφονται. Γιατί οι αγρότε αυτοί τι χάνουν διαφορετικής αντιμετώπισης από ότι οι υπόλοιποι δεν μπορώ να καταλάβω. Ο κύριος Αγνιού. Ήταν ε, πολύ καλή αυτή η επισκόπηση από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε τρεις λέξεις ε, μπορούμε να το συνοψίσουμε. Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Καταλαβαίνω τι γίνεται στην Ιρλανδία. Καταλαβαίνω γιατί καλλιεργούν και ζετάρι. Περιτοριακό να το πω και στο κύριο Φλάναγκαν και στην κυρία Μαγκίνες. Έχουμε ένα έτσι υγρό καλοκαίρι και προχαλούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Τελικά εγώ θα σας έλεγα να καλλιεργείτε κρυθάρι, το οποίο αντέχει στο χειμώνα. Πρέπει να σας πω ότι Και εμεί είχαμε θέματα με τον καιρό τα τελευταία δέκα εβδομάδα. Ε, ήταν τέλεια τα πράγματα και έχουμε πολύ καλέ σοδειέ. Έχουμε και άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε ένα ζυζάνιο το οποίο μας ε, και κάθε χρονιά, μπλακράς το ονομάζουμε, ε, κάθε χρονιά το αντιμετωπίζουμε και ο καιρός προκαλεί ανησυχίες στους αγρότες και στην Αγγλία πραγματικά αυτό που μας καίει είναι το black Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους συντονιστές που το έβαλαν στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα. Το μήνυμα από την Κομισιόν είναι σαφές ότι θα πούμε στους αγρότες ότι δεν θα υπάρξει στήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Ο λόγος είναι αυτό που είπε και ο Ιρλανδός ο Υπουργός στο Κοινοβούλιο μας που είπε ότι δεν υπάρχει ευθύνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι Ούγγροι, οι Γάλλοι όλοι αυτοί λένε ότι υπάρχει στον κλάδο κρίση. Γιατί δεν ανταποκρίνεται λοιπόν η Επιτροπή, όπως το είπε και ο Υπουργός, δεν είναι δραστήριες οι κυβερνήσεις. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις πρέπει να το κάνουν ενώ υπάρχουν οι οργανώσεις των αγροτών, υπάρχουν οι ευρωβουλευτές οι οποίοι έχουν τις ε, εκλογικές τους περιφέρειες. Υπάρχει κρίση και πρέπει να τη στηρίξετε. Υπάρχει κρίση, υπάρχει αστάθεια στις τιμές, ιδιαίτερα στη Δυτική Ιρλανδία. Δεν έχει σημασία τι τιμή θα πάρουν στην αγορά. Το προϊόν τους έχει καταστραφεί είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήταν η γαλακτοπαραγωγή, η παραγωγή κρέατος όταν οι δικοί τους τομείς ήταν σε κρίση. Η Επιτροπή λοιπόν δεν θα κάνει τίποτα. Είπατε ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλη. Αν η Ιρλανδική κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση αποφάσιζε ότι θα δώσει πληρωμή στους αγρότες για τις απώλειές τους εξαιτίας πλημμυρών ή οτιδήποτε άλλο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε ένσταση σε αυτό, θα το κατήγγειλε, γιατί εμείς εκπροσωπούμε τους αγρότες και αυτοί έχουν καταστραφεί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω φυσικά να ευχαριστήσω και εγώ και την κυρία Μαγκίνες. Κοιτάξτε, κάθε μήνα κάνουμε τη διαδρομή Στρασβούργο-Βρυξέλλες με το τρένο, πολλοί από εμά και έχουμε δει ποια είναι η κατάσταση. Υδρογραφικά στη Γαλλία, από το Στρασβούργο στη Λίλ, οι πλημμύρες ήταν φοβερές, ήμασταν με τα πόδια στο νερό. Η κατάσταση είναι τόσο τραγική που στη Γαλλία δεν είμαστε σίγουροι ότι φέτος θα έχουμε αρκετούς ε, σπόρους ποιότητας για να κάνουμε ψωμί. Τα πράγματα είναι πολύ τεταμένα. Και για να απαντήσω για το τι έγινε στη Γαλλία, αν και ο κύριος Αντρέ είναι περισσότερο καλύτερα σε θέση να το κάνει αυτό, είναι για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση των δανείων και να υπάρξει εγγύηση για ένα τμήμα βάσει μιας ε, γαλλικής δημόσιας δομής. Βοήθεια στο κεφάλαιο είναι από άλλες πηγές. Οπότε τίθεται το πρόβλημα όχι τόσο των ασφαλίσεων, γιατί αυτές δεν έχουν προβλεφθεί στην ε, ΚΑΠ, αλλά για το πώς θα χρησιμοποιηθούν ε, ταμεία αμοιβοποίησης και πού θα βάλουμε το κριτήριο, τον πύχη, για να ενεργοποιηθούν τα κονδύλια από τα ταμεία αυτά. Οι απώλειες είναι πολύ ψηλές, οπότε δεν θα είναι αποτελεσματικό το μέτρο και ίσως θα χρειαζόταν να λειτουργήσει πραγματογνωμοσύνη ώστε βοήθειες να είναι λειτουργικές. Παρακαλώ. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ που οργανώσαμε την παρουσίαση αυτή και ευχαριστώ πολύ και την κυρία Μαγκίνης που σκέφτηκαν τους Γάλλους αγρότες που υποφέρουν όπως και άλλοι εξάλλου. Είμαι παραγωγό δημητριακών αλλά και από περιοχή με πάρα πολλά δημητριακά που είναι βολόνα τη Γαλλία. Είμαστε στο κόκκινο. Όλοι έχουν 30% για τα δημητριακά πόλα, 40% για την κόλτσα, κράμβι, και 20% των Γάλλων αγροτών δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τις γεωργικές τους δραστηριότητες από τώρα, από το 2016 για το σκληρό σύτο. 65% έχουμε απώλειες σε σχέση με τους μέσους όρους 2011-2015. Με σοκάρουν αυτά που άκουσα από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που τόλμησε να πει ότι ε, πιστεύει ότι θα τα καταφέρουν οι παραγωγοί Δημητριακών της Γαλλίας. Μα πήγαινε καλά, ε, λέει, ε όχι. 50% με τα προβλήματα που έχουν με τα παριστοκτόνα, λοιπάσματα κλπ. Αν είχατε επισκεφτεί τη Γαλλία θα τα γνωρίζατε όλα αυτά. Είναι σκανδαλώδες. θυμίζω επίσης 220 ευρώ δύναμε, ενώ τώρα δίνουμε 140 μόνο ε, πληρώνουμε τους αγρότες για το σκληροσύτο. Και σε όλα αυτά φταίει η μεταρρύθμιση της κοινή λογικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να επιτρέψει στις χώρες μέλη να προστατεύσουν τους παραγωγούς τους και την παραγωγή τους και να αρχίσουμε να επανερχόμεθα στις ελάχιστες ε, ε, τιμές εγγύησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από αυτά που είπε ο κύριος Λαζό, να έχει δίκιο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το κλίμα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα κριτήρια, όμως είναι πολύ σοβαρή κατάσταση και δεν είναι δυνατόν το θέμα αυτό να το παίρνουμε έτσι στελαφιά. Πιστεύω ότι η περιγραφή της κατάστασης είναι ενδιαφέρουσα και μας υποχρεώνει να σταθούμε πάνω σε αυτή. Δεν θέλω να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριο Νταντάν. Τα εξήγησε, εξήγησε τι διαδικασίε κατεπήγοντο τη γαλλική κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Ένα τμήμα της Ευρώπης επλήγει όσον αφορά τα δημητριακά και μεταξύ άλλων η Γαλλία βρίσκονται σε πολύ μεγάλη δυσκολία. Πώς διαχειριζόμαστε λοιπόν τα εργαλεία που διαθέτουμε στην αγορά. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα μέσα στους επόμενους μήνες. Και μετά, για μετά το 2020 πρέπει να είμαστε σε θέση να προκαταλαμβάνουμε, να έχουμε δηλαδή στη διαθεσή μας τα κατάλληλα εργαλεία. Και όσον αφορά την έκθεση για την αστάθεια των τιμών, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη προσοχή για το τι θα κάνουμε στο μέλλον. Πρόκειται για τη ρύθμιση. Και από αυτού πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και να προλαμβάνουμε τις καταστάσεις. Να μην είμαστε δογματικοί, αλλά να προσφέρουμε στους αγρότες μεικτά εργαλεία ρύθμισης για να μπορούν να διαχειρίζονται την κατάσταση όσο γίνεται πιο γρήγορα για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Ευχαριστούμε. Λέει ο Πρόεδρος. Καλωσορίζουμε τους προσκεκλημένους μας. Του κύριου Νίκολσον προσκεκλημένοι είναι. Πρόκειται για φοιτητέ. Και να ξέρετε ότι χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Είμαι πεπισμένος ότι θα έχετε μια καλή εντύπωση για τη συζήτηση που κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να επανέλθω κάπως ε, σύντομα για αυτά που είπε ο συνάδελφο Φρανσίς, όχι, συγγνώμη, Ερικ Αντρία. Λέω προσοχή σε όλους μας για την αναγκαιότητα που μας υποχρεώνει και που είναι πολύπλευρη και έτσι πρέπει να δούμε αυτή την κρίση. είναι η κατάσταση που μας υποχρεώνει να κάνουμε προτάσεις οι οποίες να επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση της αστάθειας τιμών. Αναφερθήκατε σε εργαλεία διαχείρισης κρίσεων. Εγώ θα έλεγα και διαχείρισης κινδύνων επίσης. Είναι συμπληρωματικά αυτά τα δύο μεταξύ τους. Βασίζομαι λοιπόν στην δικιά σας ικανότητα να μας ακούσετε όλους ώστε να προσφέρουμε στους Ευρωπαίους αγρότες και πιο συγκεκριμένα τους Γάλλους και να προσφέρουμε λοιπόν λύσεις οι οποίες θα τους βοηθήσουν να έχουν ένα καλύτερο μέλλον και να έχουν έτσι τη δυνατότητα να αφήσουν τις ε, μονάδες τους, τις εκμεταλλεύσεις τους στην επόμενη γενιά. Κυρία Νόχη, νομίζω ότι σίγουρα στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε πολλές κρίσεις έγινε και η ακρόαση για το θέμα της αλλαγής του κλίματος πρόσφατα και νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε, πώς θα πρέπει να προετοιμαστεί η γεωργία για να μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον με την αλλαγή του κλίματος, αλλαγή της θερμοκρασίας, αλλαγή των υδάτινων συμπεριφορών. Και είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν εκ των προτέρων στρατηγικές για να αντιμετωπιστεί η αλλαγή του κλίματος και ενδεχομένω να αξιοποιηθεί και να αλλάξουν ίσως και κάποιες συμπεριφορές. Γι' αυτό λοιπόν θα υπάρξει και μία έκθεση πρωτοβουλία για το θέμα της πολιτικής ε, για τη γεωργική ανάπτυξη στην Ευρώπη και τη αντιμετώπιση ε, τη αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τι δυνατότητες υπάρχουν και να είμαστε σε ηγετικό ρόλο και όχι μόνοι να τρέχουμε τελευταία και κατεδρομένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χόιμπους. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου τύχη που μιλώ μετά την κυρία Νόεχλ, γιατί θα ήθελα να την υποστηρίξω στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν τα συστήματα καλλιεργιά μας, πώς μπορούν να δημορφωθούν με πιο ανθεκτικό τρόπο για να αντιμετωπίσουν την αλλαγή του κλίματος, τι πλημμύρε, την ξηρασία. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την ε, σύνθεση του εδάφου την περιεκτικότητα σε διάφορα στοιχεία και συμφωνώ απόλυτα, θα πρέπει να είμαστε ενεργοί και να προετοιμαστούμε. Γιατί στο μέλλον θα πληθούν όλοι οι τομεί από την αλλαγή του κλίματο και κάθε μήνα θα κάνουμε συζητήσει όπω η σημερινή. Θα πρέπει λοιπόν να επιτύξουμε ηγετικό ρόλο και να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και πιστεύω ότι αυτό αποτελεί κάθε εικόνα του Κοινοβουλίου, μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος και έτσι ολοκληρώθηκε ο κατάλογο των ομιλητών και έτσι θα μπορούσαμε να δώσουμε το λόγο εκ νέου στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή, τον κύριο Κροστέ, για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ετέθησαν και στα σχόλια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, νομίζω ότι θα πρέπει να διευκρινίσω ότι εγώ βρίσκομαι εδώ για να κάνω μια παρουσίαση για το πώ εμεί αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και πώ την ε, παρατηρούμε και την καταγράφουμε την κατάσταση στην ομέα των Δημητριακών. Νομίζω ότι σα παρουσίασα από πλευρά των εμπειρογνωμών πόσο οδυνηρή ήταν η κατάσταση σε κάποια μέρη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο ευνοϊκή σε κάποιε άλλε χώρε. συνολικά δηλαδή συνολικά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω πόσο επλήκτησαν κάποιοι άνθρωποι, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και τι μέτρα θα απαιτούνταν. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω το εξή. Πάντα το έλεγα και θα το επαναλάβω ότι τα γεγονότα τα οποία είδαμε και στον τομέα των, ε, της εκτροφής και στον τομέα των γαλακτοκομικών θα πρέπει να μας ε, προετοιμάσουν για το μέλλον, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Όπως είπε η κυρία Τελαέ, φυσικά θα τα εξετάσουμε όλα αυτά, φυσικά και θα ενημερωθούμε και θα τα λάβουμε υπόψη και για τη μελλοντική κατάρτιση, κατάρτιση της πολιτικής μας. Για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ σε ό,τι αφορά τις λύσεις κρατικών ενισχύσεων, προφανώς υπάρχουν ανέφερα το γαλλικό σύστημα. Δεν γνωρίζω να έχει ακολουθήσει κάποια τέτοια οδό κάποιο άλλο κράτο μέλο, αλλά ασφαλώ αποτελεί αυτό μία δυνατότητα και να υποενθυμίζουμε ασφαλώ τα κράτη-μέλη ότι πρόκειται για το δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ σταθεροποίηση εισοδημάτων, όπου υπάρχουν πολύ πιο πολλές και πολύ πιο εύκολες δυνατότητες υποστήριξης των αγροτών μέσω της ρυθμίσης Omnibus. Και φυσικά και την απαιτητά μέσω ιδιωτικών ασφαλίσεων οι αγρότες. Εξ όσων καταλαβαίνω, φυσικά αυτό είναι πάντα απλό. Προσπάθησα επίσης να βάλω το πολύ κακό έτος του 2016 στο συγκείμενο των προηγούμενων ετών που ήταν πολύ καλά. Και αυτό εξηγεί γιατί, για παράδειγμα, στην Ιρλανδία γίνεται τόσο μεγάλη καλλιέργεια δημητριακών, γιατί ήταν πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα έτη. Είναι σημαντική η διαφορά, θεωρώ, μεταξύ των δημητριακών των συντηρών σε σχέση με τον τομέα των γαλακτοκομικών, τον τομέα της εκτροφής ζώων, όπου βλέπουμε διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία ανακύπτουν ξανά και ξανά και προσπαθούμε κάπως να τα επιλύσουμε. Δεν πιστεύω κι εγώ ότι θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα στα δημητριακά σας σιτηρά, γιατί υπάρχει μεγάλη δραστηριοποίηση των μελών. Και η κρατική επιτροπή πάντα προσπαθεί να καταλήξει σε μια δική της τοποθέτηση τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τον χαρακτήρα των συγκεκριμένο του κλάδου αυτού των ε, σιτηρών. Καταρχάς, τα σιτηρά μπορούν να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν, να χρησιμοποιηθούν για βιοκαύσιμα. Άρα, υπάρχουν πολλές δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησης του. Φυσικά, υπάρχουν και μειονεκτήματα και θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο ασφάλειας. Η παραγωγή σιτηρών επηρεάζεται άμεσα και τις δραστηριότητες των ε, εκτροφέων ζώων. Άρα θα χρειαστεί μια συζήτηση εις βάθος για τις δυνατότητες σταθεροποίησης της κατάστασης στην πρώτη φάση της δραστηριότητας αυτής σε ό,τι αφορά την παραγωγή σιτηρών. Και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο θέμα της εμπειρίας διαταξής, αγαπητοί συνάδελφοι ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Όγκαν ο οποίος ε, και μόλις κατέφτασε και μπαίνει στην αίθουσα. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν και να τον καλέσουμε να έλθει εδώ μπροστά στο βήμα. Βλέπω πάρα πολύ θέλουν ήδη το λόγο. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός. Πολλοί κόσμος θέλει να παρέμβει. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Τι να κάνω καταρχήν, να δώσω το λόγο στον Επίτροπο ή να δώσω το λόγο σε εσά. Όχι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Θα ξεκινήσουμε ως ήθιστε. Ας πω εγώ, καταρχάς, κάποια εισαγωγικά λόγια. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω πολύ. Θα πω λίγα λόγια και θα περάσουμε αμέσως μετά στην παρέμβαση του Επιτρόπου. Για να μην πω ότι θα πρέπει, επειδή έχουμε τόσες ερωτήσεις, κατηγισμό ερωτήσεων, να δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να ακούσουμε και εσάς. Λοιπόν, θέλουμε να μιλήσουμε για την πρόταση Omnibus για τη γενική πρόταση αυτή έρχεστε την κατάλληλη στιγμή γιατί έχουμε και, την, και τον πρόεδρο εδώ της Επιτροπής Προπολογισμών που, ήταν, που είναι και ένα πληρωματικό μέλος της δικής μας Επιτροπής. Χαιρόμαστε που είστε εδώ κύριε Πρόεδρε και ξέρω τα γεωργικά θέματα ότι είναι πολύ σημαντικά για σας. Καλώς ήρθατε. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές. Χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω να μιλήσω στην Επιτροπή σας για να παρουσιάσω την πρόταση της Κομισιόν, τη λεγόμενη πρόταση Omnibus που υιοθετήθηκε τον περασμένο μήνα από την Επιτροπή. Ε, λογικό είναι να συζητήσουμε σήμερα, γιατί τη Δευτέρα το συζητήσουμε αυτό το θέμα με το Συμβούλιο των ε, Υπουργών. Ε, θα ακούσουμε μια πρώτη αντίδραση των Υπουργών ε, στα διάφορα μέτρα που προτείνουμε. Υπάρχουν διάφορα θέματα που θα ήθελα να σταθώ στην παρουσίασή μου ε, και θέλω να τη θέσω στο σωστό πλαίσιο. Ε, είναι τμήμα της ενδιάμεσης έκθεσης, μια και βρισκόμαστε στα ενδιάμεσα της περίοδου χρηματοδότησης. Ε, ξέρω ότι το θέμα αυτό σα απασχολεί και εσά όπω και το Συμβούλιο. Και τέλο θέλω να πω και κάποιο από το περιεχόμενο που σχετίζεται με τι βασικέ αλλαγέ και, τους, ε, και αυτές οι αλλαγές αφορούν τους τέσσερις κανονισμούς της ΚΑΠ. Ε, την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε ε, αλλά όχι σε υπόθεμα χαρτιού η πρόταση αυτή, ε, με τι αλλαγέ στους τέσσερι κανονισμού, το πλαίσιο γιατί προτείναμε αυτές τις αλλαγές κτλ. Ο κανονισμό Omnibus είναι βασικό τμήμα τη ενδιάμεση έκθεση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Η ενδιάμεση έκθεση ήταν τμήμα τη Πολιτική Συμφωνία για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ο στόχος της Κομισιόν ήταν να πλουστεύσει του κανόνες, επί των οποίων τα κράτη-μέλη και άλλοι δικαιούχοι λαμβάνουν τα χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προτινόμενη απλούστευση των κανόνων αφορά διάφορους κανόνες και θα έχει διάφορα αποτελέσματα. Θα έχει ευκολότερη πρόσβαση στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενθαρρύνει τους πολίτες ε, να ε, ξοδεύουν σωστά τα χρήματα, θα έχουμε μείωση κατά 25% ε, στο, στο, ποσό, στο ποσό αυτό. Οι προτάσεις του Omnibus είναι ουσιαστικές ε, και αφορούν την ατζέντα πλούστευσης. Θέλουμε να εντοπίσουμε διάφορα μέτρα, ούτω ώστε να έχουμε πολιτική επιτυχία χωρίς να αλλάξουμε όμως τους προσανατολισμούς. Το, καμία ουσιαστικά πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό διάφορα μέτρα τα οποία ε, θα θέλατε να συμπεριληφθούν, ίσως δεν έχουν συμπεριληφθεί τελικά στο Omnibus. Ξέρω πολύ καλά ότι η εμπλοκή της Επιτροπής σας στην ε, νομοθετική διαδικασία ε, είναι πολύ έντονη. Γιατί είναι σημαντικό αυτό το θέμα για σας. Και μετά τη συνάντηση με τους ε, υπουργούς τη Δευτέρα, ε, θα δείτε την έκθεση, θα δείτε και την έκθεση του Συμβουλίου και θα δείτε και τις επιφυλάξεις των Υπουργών για την νομοθετική διαδικασία. Να επαναλάβω αυτό που έχω πει ήδη στο Συμβούλιο, ότι η πρόταση της Κομισιόν έχει οθετηθεί και θα πρέπει όμως να συμφωνήσουν τώρα οι συνομοθέτες ε, θέλουμε να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, να εξασφαλίσουμε την ε, συμφωνία. Ε, στα περισσότερα στοιχεία του πακέτου ή δυνατόν αυτό το τέλος του 2016, τόσο ώστε να τεθεί σε ισχύ 1η Ιανουαρίου του 2018. Να ισχύσει δηλαδή για τα τελευταία τρία χρόνια του τρέχοντος πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ε, το είπα στο Συμβούλιο και διάβασα και τις εκθέσεις ε, τις δικές σας για τη διαδικασία. Θέλω να σα ξεκαθαρίσω, ο Κομισιόν ε, δεν υπαγορεύει το πώς ε, οι άλλοι θεσμοί λειτουργούν στο εσωτερικό τους. Η... Θέλουμε απλώ να βοηθήσουμε στην όλη διαδικασία, ώστε να φτάσουμε σε μια διαθεσμική συμφωνία για μια πλειάδα μέτρων, τα οποία καταρχά θα υποφεληθούν, από τα οποία θα υποφεληθούν κυρίω οι γεωργοί μα. Θα είμαι επικοδομητικό, θα συνεργαστώ και εγώ και οι υπηρεσίε μου ε, υπό οποιαδήποτε μορφή ε, χρειαστεί στα πλαίσια τη νομοθετική διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω Ε, με αυτόν τον τρόπο να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία. Η πρόταση Omnibus Κομισιόν έχει μία σειρά από τεχνικέ αλλαγέ στου τέσσερι βασικού κανονισμούς τη ΚΑΠ. Για την ανάπτυξη υπαίθρου, για την ΚΟΑ, τον οριζόντιο κανονισμό και τον κανονισμό για τι άμεσες πληρωμές. Αυτές οι προτινόμενε αλλαγέ μετά την ε, εκτενή εξέταση της νομοθεσίας που έγινε πέρυσι ε, καλύπτουν την απλούστευση, την ευελιξία και την επικουρικότητα. Η ιδέα ήταν το Omnibus να έχει διάφορα μέτρα απλούστευσης, τα οποία δεν θα αλλάζουν τους γενικούς προσανατολισμούς της πολιτικής. Αυτή ήταν η προσέγγιση μου, συνεισφέροντας την πρόταση της Κομισιόν. Ε, επομένως, περιορίστηκα σε, στα προβλήματα, εκεί που είχαμε κόλλημα, εκεί που είχε πρόβλημα και, είχαν πρόβλημα και τα κράτη-μέλη και η Γεωργία και οι αρχές πληρωμής. Επίσης, ε, πολλά από τα μέτρα είναι πολύ φύσεω, φύσεως, μια και αφορούν πληρωμέ. Θέλω να εστιάσω στα μέτρα τα οποία θα εξασφαλίσουν μια απλούστευση της ΚΑΠ. Εκεί εστίασα. Ε, για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Έχουμε μια τομεακή διάταξη για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων. Θα έχουν τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν ε, εργαλεία τα οποία θα είναι, συγκεκριμένα για, ε, θα είναι συγκεκριμένα για κάποιο τομέα, που θα είναι πιο ελκυστικά και για τις διοικήσεις και για τους γεωργούς. Ε, Ούτω ώστε να έχουμε καλύτερα μέσα ε, για να στηρίξουμε τους γεωργούς σε περιπτώσεις κρίσης, και μην ξεχνάτε ότι οι, διαφο οι εμπειρίες είναι τελείως διαφορετικές από τομέα σε τομέα. Επομένως, αυτή η αλλαγή μπορεί να ανταποκριθεί ε, στην αντιμετώπιση των κρίσεων σε κάποιες γεωργικές αγορές. Επίσης, θα πρέπει ε, να δούμε κατά πόσο υπάρχει η συμμόρφωση με τα μέτρα ΠΟΕ, ε, αυτού του μέτρου δηλαδή και του ΠΟΕ. Ε, Έχουμε το Amber Box και εκεί εμπίπτει στα πλαίσια του ΠΟΕ, ε, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει αρκετό περιθώριο για να περάσουμε αυτό το μέτρο. Μια άλλη αλλαγή είναι απλούστεροι κανόνε για την πρόσβαση των, ε, σε δάνεια και σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ούτω ώστε να χρησιμοποιούμε καλύτερα στο γεωργικό τομέα τα χρηματοδοτικά μέσα να έχουμε καλύτερη ε, πρόσβαση σε κεφάλαιο για γεωργούς, κυρίως νέους αργογούς, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με την πίστοση η πρόταση ε, ανταποκρίνεται στις ανησυχίες που έχουν ε, εκφράσει διάφοροι σε ό,τι αφορά τη, τη γεωγραφία, ε, την γραφειοκρατία, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην πίστη. Θέλουμε να ενθαρρύσουμε καλύτερη μόχλευση του δημοσίου χρήματος και να υπάρχει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στη γεωργία. Ε, θα έχουμε τη δυνατότητα να κινητοποιήσουμε περισσότερα ποσά μέσω των επιχορηγήσεων. Ε, και θα υπάρχει και δυνατότητα επαναχρησιμοποίηση τους στο μέλλον. Επιτέλους θα έχουμε και απλούστερους κανόνες για τους νέους γεωργούς. Ε, τα κριτήρια επιλογής αλλάζουν, ούτω ώστε και η ζωή των αρχών, των αρμοδίων αρχών να είναι πιο εύκολη. Άμεσες πληρωμές. Αλλαγέ έχουμε εκεί, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν εάν θέλουν να συνεχίσουν ή όχι ε, να εφαρμόσουν τον ορισμό του ενεργού γεωργού. Εάν ναι, το σύστημα θα γίνει πολύ λιγότερο ε, επαχθές, ας πούμε, και θα μειωθεί και το κόστος και για τους γεωργούς και για την, ε, ε τις διοικήσεις. Ε, εδώ είχαμε πολλές αντιδράσεις στο Συμβούλιο από κρατημέλη γιατί συμφωνούμε αυτή την ευελιξία που εισάκουμε. Ενώ κάποιοι εξέφρασαν και ανησυχία για την επίπτωση που θα έχει, ε, μήπως δηλαδή δημιουργήσει ε, μη ίσους όρους ε, ανάμεσα στους δικαιούχους και μη δικαιούχους. Λοιπόν, πέρα από το θέμα τη ε, ευελιξία, οποιοδήποτε φορέα λαμβάνει άμεση στήριξη θα πρέπει να συμμορφώνεται με τον ορισμό του γεωργού. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιο να ασκεί γεωργική δραστηριότητα σε γεωργική γη. Ε, αυτή η σημαντική διευκρίνηση πιστεύω ότι θα διασκεδάσει κάποιε από τι ανησυχίε που είχατε σε ό,τι αφορά του νέου γεωργού. Η πρόταση θα εξασφαλίσει ότι το ποσό του 2% ξοδεύεται πλήρω χρησιμοποιώντα ε, το μέγιστο ποσό εκταρίων μόνο αν τα ποσά ε, δεν επαρκούν για να καταβληθούν, τα ποσά δεν αρκούν για όλες τις ανάγκες. Επίσης, έχουμε αλλαγές για τα SAPS και την ε, συνδεδεμένη ενίσχυση, ούτως ώστε να χρησιμοποιούνται καλύτερα αυτά τα κονδύλια. Σε σχέση με την εθελοντική συνδεδεμένη ενίσχυση, η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει την δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν να δίνουν και αποσυνδεδεμένη βοήθεια με βάση τις παλιές ιστορικές περιόδους για μεγαλύτερη περίοδο από 12 μήνες. Ο στόχος του μέτρου είναι να μπορούν οι γεωργοί να λαμβάνουν τα ίδια ποσά συνδεδεμένης βοήθειας χωρίς ε, να, έχουν τον, να πρέπει να κρατήσουν τον ίδιο αριθμό ε, παραγωγικών μονάδων. Θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη ε, που έχουν λιγότερους παραγωγούς ε, στα προκυπευτικά να αυξήσουν την ε, στήριξη στις οργανώσεις παραγωγών χωρίς να υποβάλουν πρόταση στην Κομισιόν κατά ανάγκη. Επιπλέον, ε, θέλουμε να βοηθήσουμε τις οργανώσεις αυτά τα κράτη-μέλη και έχουμε την, λεγόμενη, το λεγόμενο coaching, δηλαδή την βοήθεια, την παροχή συμβουλών ας πούμε, στους, στις οργανώσεις. οι νέες ειδικά οργανώσεις μπορούν να υποφεληθούν από την εμπειρία ή από την εμπειρία που έχουν οι πιο παλιές οργανώσεις. Τέλος, Πρόεδρε, στον οριζόντιο κανονισμό ε, έχουμε πιο αναλογικούς κανόνες για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και επίση για την διόρθωση των παρατυπιών. Ε, επίση, μια προστατευμένη διαδικασία για τη διαχείριση τη δημοσιονομική πειθαρχια πειθαρχίας. Διάφορα κράτη-μέλη εξέφρασαν ανησυχίες για την πρόταση να αντικαταστήσουμε τον κανόνα 50-50 με έναν απλό κανόνα εκαθάριση 100%. Αλλά μερικέ χώρε δεν κατάλαβαν ότι αυτή η πρόταση είναι μια μεγάλη απλούστευση και για τα κράτη-μέλη και για την Κομισιόν. Παράλληλα, ανταποκρινόμαστε στις επικρίσεις ε, της ε, επιτροπή σα. Τη αρμόδια Επίτροπή, ότι χρειάζεται ε, τεράστιο χρονικό διάστημα για να ανακτήσουμε το υπόλοιπο 50% α πούμε. Η δημοσιονομική επίπτωση ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι πολύ λίγο. 17 ε, μέχρι 22 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία τρία χρόνια. Τα κράτη-μέλη θα έχουν μικρότερο γραφειοκρατικό άχθο. και τα παράνομα ε, δάνεια ε, θα μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να τα διεκπαιρεώνουν πολύ πιο εύκολα, γιατί δεν θα πρέπει να καταβάλουν τόσες πολλές αποδείξεις. Κύριε Πρόεδρε, ε, επίσης μου ζητάτε να επιταχύνω την απλούστευση. Ο, το Omnibus είναι ένα βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ε, μπόρεσα χάρη στο Omnibus να προτείνω βασικές αλλαγές στις βασικές πράξεις. Το Omnibus δηλαδή είναι μια πρόταση που θέλει να διασκεδάσει, να εξαλείψει διάφορα προβλήματα ε, υπέρ του Γιώργου τελικά. Εκτιμώ ότι κι εσείς όπως και πολλοί υπουργοί Μπορεί να έχετε επιφυλάξει για τη διαδικασία. Εξήγησα όμω τη θέση τη Κομισιόν γι' αυτό και σα διαβεβαιώ ότι είμαι διατεθειμένο να συνεργαστώ με οποιαδήποτε μορφή προτιμάτε εσεί, ούτω ώστε να, ε, να τελεσφορήσει αυτή η πρωτοβουλία. Θα πρέπει βεβαίω να ληφθεί απόφαση με συναπόφαση εδώ, ε, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο. Επίση, σήμερα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μια αρχική ανταλλαγή απόψεων για όλα όσα λέει αυτή η πρόταση να ακούσετε τις προτάσεις μου και να ακούσω κι εγώ τις πρώτε αντιδράσεις. Βεβαίω, χωρίς να προδικάζουμε την όποια θέση θα πάρει το δικό σας θεσμικό όργανο ή τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα σε μεταγενέστερη φάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε πίτροπε. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους συντονιστές, δύο λεπτά ο καθένας. Και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους ευρωβουλευτές, ένα λεπτό καθένας. Ο κύριος Ντες πρώτα. Δύο λεπτά παρακαλώ κύριε Ντες. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε και τον Επιτρόπο Χόγκαν που βρίσκεται μαζί μας στην Επιτροπή αγροτική ανάπτυξη και μας παρουσιάζει την πρόταση Omnibus. Ε, ήμασταν υπόμονοι και περίεργοι όλοι και η ομάδα μα σίγουρα θα συνεργαστεί μαζί σας προκειμένου να σταθούν με επιτυχία αυτέ οι προτάσει. Μίλησατε για μια μεγάλη σειρά προτάσεων απλοποίηση. Νομίζω ότι θα είσαστε ο πρώτος επιτροπός που θα πετύχει να υπάρξει όντω απλοποίηση, αν το πετύχετε. Γιατί συχνά μιλάμε για απλοποίηση στην πολιτική, αλλά συνήθω αυτό προκαλεί πιο πολύ η γραφειοκρατία. Τώρα λοιπόν έχουμε επιτέλου την ευκαιρία πραγματικά να πλουστεύσουμε μια διαδικασία. Το περιμένουν με ανυπομονησία αυτό οι αγρότε μα. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιδείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα. Το πιο σημαντικό λοιπόν θέμα για μα, και αυτό είναι αυτονόητο θεωρούμε, είναι να υπάρξει η κατανομή, η διέρεση της ε, νομοθεσίας Omnibus. Λοιπόν, νομίζω ότι θα πρέπει να βγάλουμε τους τέσσερις τροχούς του οχήματος Omnibus και να τις ε, δώσουμε τον καθένα στην αρμόδια επιτροπή. Θα πρέπει να το εκφράσουμε αυτό. Δεν έχουμε οποιαδήποτε δυσπιστία προς την Επιτροπή του προπολογισμού. Έχουμε εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα για τις προτάσεις αυτές και θα πρέπει πλέον λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και νομίζω ότι αυτό μας βρίσκει σύμφωνο ε, από όλες τις ομάδες και θα ήθελα να κάνετε κάποια παρατήρηση κατά πόσον υποστηρίζουν υποστηρίζετε αυτή την πρότασή μας. Νομίζω ότι το Συμβούλιο θα έχει παρόμοιες θέσεις για το θέμα αυτό και αν θα μπορούσαμε να τα κοιτάξουμε αυτά από κοινού, νομίζω το αποτέλεσμα θα είναι καλό. Τελευταία παρατηρήση στις ε, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Θα θέλαμε να σας ε, παρακαλέσουμε να μην προκληθούν, να μην προκύψουν αυτές οι 15 εκτελεστικές πράξεις από μία μόνο εκτελεστική πράξη, αλλά να τις ψηφίσουμε ξεχωριστά. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και θα συνεργαστούμε σίγουρα μαζί σας προκειμένου να υπάρξει επιτυχημένη έκβαση. Ο κ. Ε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Φυσικά, εμείς συμφωνούμε με αυτή την ε, προσέγγιση για την ε, απλούστευση. Ελπίζουμε ότι αυτή η πρόταση θα έχει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν θα μπω στην ουσία, Φυσικά οι τίτλοι που μας αναφέρατε είναι πολύ ενδιαφέροντες. Μεγάλη ευελιξία, ε, νέοι, σταθερό εισόδημα. Όμως, Επίτροπε, αυτό που μας ανησυχεί είναι η διαδικασία που επιλέξατε. Αυτή η διαδικασία Omnibus κινδυνεύει πραγματικά και το τονίζω, γιατί τα είπαμε εδώ μεταξύ μας, εδώ στην Επιτροπή. Ε, το πρόβλημα δεν είναι η έκθεση που θα προκύψει από την Επιτροπή μας, εδώ, η δική μας έκθεση, δηλαδή η κοινοβουλευτική. Το θέμα είναι τι γίνεται στις ε, διαπραγματεύσεις, ε, στους τριμμένους διαλόγους. Εμείς ως Επιτροπή Γεωργίας ε, κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε άλλο στρατόπεδο, να πρέπει να διαπραγματευτούμε με ποιον, με το ΕΚΟΦΗΝ, με τον Επίτροπο Υπεύθυνο για τον Προϋπολογισμό. Εμείς μας, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να βγουν αυτοί οι τέσσερις βασικοί κανονισμοί από το πακέτο Omnibus. Έτσι. Και αυτό δεν είναι σπατάλη χρόνου. Εγώ είμαι ο, ε, ο γενικός εισηγητής και έχω από κάτω μου 7 υποεισηγητές όπου εξετάζουμε τα θέματα της αλληλείας, της ε, περιφερειακής πολιτικής κτλ. κτλ. Όλες τις πολιτικές. Προσπαθούμε δηλαδή να συνεργαστούμε όλοι μας. Και γράψαμε και στον πρόεδρο της διάσκεψης των προέδρων. Πρέπει να δούμε το θέμα της διαδικασίας, της διαπραγμάτευσης, γιατί αλλιώς αντί να πλουστεύσουμε τα πράγματα θα τα περιπλέξουμε. Ελπίζω να, μας, να μπορέσετε να μας βοηθήσετε λιγάκι με το θέμα της διαδικασίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω τον Επίτροπο στην Επιτροπή μας. Δεν τον εκπλήσει το ότι το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας αυτό το θέμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσω εδώ ότι βεβαίω και θέλω την αρχή της απλοποίησης και καλωσορίζω τις προσπάθειες που έχουν γίνει επί τη ουσίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολλές από τις ανησυχίες των μελών της Επιτροπής Γεωργίας αλλά και από τους ίδιους τους γεωργούς. Σε σχέση με τους νέους αγρότες, η σταθεροποίηση του εισοδήματο, για παράδειγμα σε διάφορους τομείς και η ανταπόκριση στις ανάγκες τους με νέα οικονομικά μέσα, όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσέ προτάσεις, αναμφίβολα η Επιτροπή μας είναι υπέρ της απλοποίησης, εννοείται. Και εκτιμούμε το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη της η Επιτροπή της Ανησυχίας μας. Όμως, ως Επιτροπή, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τον τρόπο με τον οποίο έχει δουλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα και έχει αποκλείσει από τις διαπραγματεύσεις τους εκπροσώπους της Επιτροπής Γεωρίας παρόλο που είμαστε συνομοθέτες. Το μήνυμα είναι ότι αν συμμετέχει η άκρη που έχει νόμιμα ε, δικαιώματα και συναποφασίζει νομοθετικά θα δυσκόλευε την διαδικασία, λέτε. Γιατί δεν θα μπορούσαμε και εμείς να βοηθήσουμε. Εμείς διαπραγματευθήκαμε και βοηθήσαμε να βρεθούν λύσεις στην αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Είναι απαράδεκτο να γίνονται αλλαγές χωρίς πλήρη διαβούλευση μαζί μας. Ξέρω ότι το θεωρεί διοικητικό ζήτημα η Επιτροπή, αλλά δεν είναι έτσι. Εμείς θα φροντίσουμε να αναλαμβάνουμε τις νομικές μας ευθύνες απέναντι στον αγροτικό κόσμο. Θα τελειώσω με το εξή. Την αναθεώρηση της ΣΚΑΠ την κάναμε, περάσαμε από αυτή τη διαδικασία. Δεν ήταν εύκολο αλλά συναποφασίζαμε, ήταν δικαίωμα της Επιτροπής μας. Δεν μπορεί τώρα να, να παρατηθούμε από ένα τέτοιο δικαίωμα, όπως το είχαμε με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και τώρα να παρετηθούμε από αυτό. Ε, ευχαριστούμε. Κυρία Μούλερ, ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονό ότι μου δίνετε το λόγο εξ ονόματο του συντονιστή μα. Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι θέλετε να προβούμε σε απλοποιήσεις και να επιλύσουμε τα προβλήματα. Φυσικά αυτό το υποστηρίζουμε. Είμαι υπέρ της απλούστευσης, αλλά νομίζω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είμαι σχετικά καινούργια και δεν έχω συνεργαστεί για την κατάρτιση ε, πράξεων κατά εξουσιοδότηση, αλλά ξέρουμε ότι από την πρακτική εμπειρία μας ότι συχνά εδώ στο Κοινοβούλιο υπάρχει αυτή η τάση να ζητάμε τέτοια συμμετοχή και είμαι λίγο απογοητευμένη που στην διαδικασία Omnibus επιλέγουμε να εισακούσουμε τις απόψεις του Κοινοβουλίου μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Χαίρομαι λοιπόν που προδίκατε στις δηλώσεις αυτές σήμερα και που θα προωθήσουμε μια ενιαία διαδικασία, αλλά θα ήθελα να προσέξουμε για την ε, κατανομή της ε, Omnibus και για τη διατηρήση της πλήρους ε, εξουσίας του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να εργαστώ για τον ορισμό των βοσκοτοπιών, για παράδειγμα, των μόνιμων αυτών ιών γιατί πρόκειται για θέματα που μας καίνε, μας απασχολούν πάρα πολύ και θα ήθελα να δούμε από κοινού το τι χρειάζεται στην πράξη. Δεν ε, υπονοώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν τα γνωρίζει αυτά, αλλά γι' αυτό μας εξέλεξαν άλλωστε. Και υπάρχουν και παιχνίδια εξουσίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής και εμείς απλά θα θέλαμε να εκφραστεί 100% και η άποψη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Σάντρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το οποίο θέλω πρώτα απ' όλα να πω είναι ότι η τροποποίηση του ορισμού ή της εφαρμογής των ορισμών για τον ενεργό αγρότη για μένα είναι πράγματα τα οποία δεν είναι απλά τεχνικά και έχουν να κάνουν με το ότι θέλετε να αλλάξετε κριτήρια τα οποία έχουμε ήδη συμφωνήσει στην κοινή γεωργική πολιτική. Η Επιτροπή μας έχει δικαίωμα λοιπόν να τα συζητήσει, να εμβαθύνει σε αυτά και να περάσουν από την Επιτροπή μας πρώτα και όχι να μπαίνουν από την πίσω πόρτα. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι, που είναι ουσίας, είναι η απόφαση δημόσιο χρήμα να πηγαίνει ενώ οι κρίσεις για τις οποίες πηγαίνει αυτό το χρήμα στους αγρότες οφείλονται σε πολιτικές αποφάσεις, όπως για παράδειγμα με το εμπάργο της Ρωσίας. Αυτά λοιπόν όλα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να περνάνε από την Επιτροπή μας. Είπατε ότι δεν είναι δικιά μας ευθύνη. Ναι, ο τρόπος με τον οποίο εσείς παρουσιάσατε τα πράγματα φταίει για το ότι δεν πέρασαν από εμά. Οπότε είναι πολύ σοβαρό αυτό. Οι ευρωβουλευτές, εμείς εδώ, εκπροσωπούμε αυτούς που μας εξέλεξαν. Και αυτοί που μας εξέλεξαν θέλουν να μπαίνουμε σε βάθος, να είμαστε αρμόδιοι και να κοιτάμε τις αλλαγές που θέλετε εσείς να επιφέρετε. Τώρα, για παράδειγμα, με το Omnibus. Είναι Επίτροπε, δεν είναι δυνατόν να μένουν απ' έξω και να μην ανακατευτούμε και εμείς βαθιά σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. ευχαριστώ. Ε, σπάνια συμφωνούμε όλες οι ομάδες εδώ στην Επιτροπή, αλλά σε αυτό συμφωνούν όλες οι ομάδες. Έτσι πώς μας το παρουσιάζετε, πολύ απλά δεν ε, είναι δυνατόν να γίνει αυτό που προτείνετε. Δεν μπορείτε να μας διαγράψετε και να διαγράψετε τις αρμοδιότητες που μας έδωσε η συνθήκη της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, αυτά που προτείνετε και στην Επιτροπή Προπολογισμού. Όλα αυτά τα πουλάτε με τον τίτλο της απλούστευσης και της απλοποίησης. Όχι, κοιτάξτε, δεν είναι θέματα, δεν είναι μόνο θέματα απλούστευσης, είναι και θέματα περιεχομένου που αλλάζουν. στοχοθέτηση, για παράδειγμα, του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά ε, τα θέματα της ουσίας δεν ε, έχουν να κάνουν με θέματα απλοποίησης και αλλάζεται για παράδειγμα τα θέματα της, ε, των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης. Μιλάτε για αλλαγές που θα σήμαιναν αλλαγή εκβάθρων του δευτεροπυλώμα. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε με αυτά ε, τυφλά. Η Επιτροπή Προπολογισμού θα εξετάσει τα θέματα δηλαδή περιεχομένου και εμεί απλά στο τέλο έρθουμε να τα κοιτάξουμε. Είναι δυνατόν να αφήσουμε να καταπατούνται τα δικαιώματά μα ω Κοινοβουλίο ανεξάρτητα από το πώς ε, τα κρίνεται όλα αυτά και από το αν λέτε ότι απλά πρόκειται για απλούστευση. Η διαδικασία που ακολουθείτε δεν ναι, είναι ανάρμοστη και είναι πραγματικά θεωρούμε προβληματικό το γεγονός ότι έρχεστε εκ των υστέρων και μας τα αναφέρετε αυτά. Γιατί το μα ενημερωθήκατε και δεν, ενημερώσετε και δεν συζητήσατε με την Επιτροπή μας εκ τον προτέρων τα ζητήματα αυτά. Και ως εκ τούτου το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν τα δεχόμαστε όλα αυτά. Εάν δεν συζητήσετε όλους τους κανονισμούς και τους τέσσερις κανονισμούς με ε, το Κοινοβούλιο πολύ απλά δεν τα δεχόμαστε όλα αυτά, γιατί πολύ απλά θα δημιουργηθεί η εντύπωση ότι υποβάλλεται δηλαδή μια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς απλά λέμε ένα ναι ή ένα ναι, όχι. Έμα έχει αλλάξει ο κόσμος από το 2009 και μετά, ξέρετε, με κρυσαγνιό. Επίτροφε, την τελευταία φορά που ήμουν στο Κόρκ στην ε, Δημοκρατία της Ιρλανδίας, μέρος που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τότε είχατε πει κάτι πολύ γενές αυτή μου εκείνο το απόγευμα που συναντηθήκαμε. Σας συγχωρώ, δεν θα το επαναλάβω τώρα. Τρία σημεία. Πρώτον, ψηφίσαμε Brexit. Πολλοί αγρότες θέλησαν να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί διαπίστωσαν ότι τους ήταν υπερβολικά περίπλοκο και δύσκολο να πάρουν τα λεφτά τους από το πρόγραμμα για το περιβάλλον. Βέβαια, αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Απ' την άλλη, μπορεί κανείς ως νέος μετανάστης να πάρει πολλά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνομαι βέβαια κοινικό εδώ. Το άλλο που θέλω να πω δεν έχει αναφερθεί καθόλου εδώ, πρόκειται για τις αγελάδες φαντάσματα. Άμα θέλετε στήριξη, ε, διάφορα βοηθή αλλά αναρωτιόμαστε υπάρχουν πράγματι εκεί ή όχι. Εσείς έχετε κάποια ιδέα για το πώς θα αντιμετωπίσετε τέτοιου είδου απάτες. Τέλος, κάποιος την Επιτροπή, ή εσείς κάποιος άλλος, δεν θέλει δεν θέλουν παριστοκτόνα στα όσπρια. Είμαστε σε τέτοια τιμή που θα μπορούσαμε στην Αγγλία να τα παράγουμε με κέρδος αλλά επειδή υπάρχουν τα πράσινα λόμπι δεν θέλουν να χρησιμοποιηθούν παρασιτοκτόνα. Και ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε σοδιές, φασόλια κτλ. που δεν θα είναι γενετικά τροποποιημένα. Εσείς κάνετε τα πράγματα πιο δύσκολα. Θα μου απαντήσετε κάποια άλλη φορά εσείς. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κάθεστε δίπλα στους ε, οικολόγους, ε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι έρχεται με όχι αποτελεσματικά μέτρα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τροποποιώντας τέσσερις βασικούς κανονισμούς. Η πρότασή σας τροποποίησης του κανονισμού για την ανάπτυξη της υπαίθρου προβλέπει απαγόρευση για διάφορα οικονομικά μέτρα υπέρ των αγροτών. Εντάξει, ο τρόπος που το βλέπετε μπορεί να είναι θετικό, αλλά δεν βλέπω εγώ καμία σχέση με την κρίση που διανύουμε σήμερα. Νομίζω ότι μια απλώς διαρθρωτική ε, παρέμβαση του αναγκάζει να εξαρτώνται πιο πολύ από τις τράπεζες. Η τιμή των αγορών είναι πολύ χαμηλή, ενώ η τιμή, το τίμα πρέπει να πληρώσω για την παραγωγή είναι πολύ ψηλό. Έπειτα για το θέμα του ενεργού αγρότη. Η κάθε χώρα, αν κατάλαβα καλά, μπορεί να αποφασίσει να συνεχίσει ή όχι να την εφαρμόζει την έννοια αυτή. Ποιο θα το κρίνει όμως. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση. Δημιουργείται διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Εμείς θέλουμε να διατηρηθεί ο ορισμός που είχαμε μέχρι τώρα για τον ενεργό αγρότη και να τηρείται παντού. Νομίζω ότι όλοι εδώ μέσα γνωρίζουμε κάποιον λιγότερο ή περισσότερο ενεργό αγρότη. Οπότε συμφωνώ με τον συνάδελφο συμφωνώ και με τον κύριο Ζωζέ Μποβέ και ξέρετε, σήμερα η αστυνομία βρέθηκε στο αεροδρόμιο. Υπάρχουν αγρότες που θεωρούνται περισσότερο ή λιγότερο λοιπόν ενεργοί. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους παραγωγούς των αγροτικών προϊόντων. Απ' την άλλη έχουμε τη ΣΕΤΑ, τη ΤΥΠΗ που θα μας οδηγήσουν σε χειρότερη κατάσταση. Καρσία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να επαναλάβω και εγώ τα ίδια, αλλά προπολογισμό. Λοιπόν, να μεταφέρουμε σε άλλες πολιτικές τα περιθώρια της ΚΑΠ είναι κάτι που το έχουμε δει στο παρελθόν και είναι πολύ κακό. Λέμε ότι τελικά, λέτε μάλλον ότι πληρώσαμε την κρίση ε, στην γαλακτοπαραγωγή από τα περιθώρια αυτά. Ωραία, γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά σε άλλες πολιτικές του κοινοτικού προπολογισμού. Τώρα για τα τεχνικά μέτρα. Λέτε να αυξηθούν τα εκτάρια για τους νέους αγρότες γιατί να μην αυξηθεί αυτό που παίρνουν όταν ξεπερνάνε το 2%. Και επειδή δεν έχω χρόνο το τελευταίο ενεργό αγρότη, είπατε ότι μετά από όσα συζητήσαμε εδώ για τον ορισμό του ενεργού αγρότη στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, τώρα γιατί θέλετε να αφήσετε αυτή την ελευθερία στις χώρες έλλη Μπορεί να οδηγήσει σε αδικίες. Ένας αγρότης ε, που βρίσκεται λίγα μέτρα από κάποιον άλλον και τους χωρίζουν σύνορα, να βρίσκονται σε δύο εντελώς διαφορετικές ε, καταστάσεις. Ο κύριος Βούδα Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ σήμερα και σας ευχαριστούμε που δέχεστε να συζητήσετε μαζί μας για την απλοποίηση της ΚΑΠ. Είναι σημαντικό Το διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα να καθόμαστε, να τα συζητάμε και να τα λύνουμε όλοι οι συνάδελφοι εδώ δεν συμφωνούν τα περιθώρια της ΠΑΚ να πηγαίνουν σε άλλες πολιτικές, ενώ στη Γεωργία δεν έχουν λυθεί ακόμα ένα σωρό, προβλήματα. Για τα τεχνικά ζητήματα τώρα. Στη Ρουμανία, όσον αφορά το νέο αγρότη, πιστεύω πως πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο σε αυτό και να στηρίξουμε περισσότερο τους συνεταιρισμούς για να μπορούν οι αγρότες να δημιουργούν τις δικές τους δυνατότητες εμπορίας των προϊόντων τους μετά την παραγωγή. Είναι σημαντικό. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με την έννοια του ενεργού αγρότη. Έχει γίνει πολλή συζήτηση, πιστεύω ότι πρέπει να τον ξαναδούμε αυτόν τον ορισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συντονιστές κι εγώ. Θέλω μια συγκεκριμένη πρόταση. Θέλω να επιστήσω την προσοχή του Επιτρόπου σε αυτό. Αν πρόκειται για επιπλέον προϋπολογισμό, συμπληρωματικό προϋπολογισμό, τότε από το 3,68 θα πάμε στο 1%. η πρόταση επίσης για τις επιστροφές με απασχολεί. Και έχει να κάνει με πολλές χώρες. Πρέπει να επανέλθουμε και γι' αυτό. Έπειτα το θέμα των ε, αδρευμένων ε, επιφανειών. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να μειωθεί. Όταν υπάρχει νερό, η δυνατότητα πρέπει να υπάρχει, έτσι κι αλλιώς. Ε, κύριε κυρία Πατήρη, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον Επιτρόπο που ήλθε εδώ σήμερα για να μιλήσει για τα θέματα απλούστευσης της ΚΑΠΑ. Όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ελπίζω ότι η απλούστευση αυτή θα επιτευχθεί. Διάβαζα λοιπόν το έγγραφό σας ε, 250 σελίδα για την απλούστευση, την απλοποίηση και θα πρέπει να σας πω ότι ειλικρινά ανησυχώ στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ξέρετε, το Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτη. και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή και να υπάρξει πραγματική απλούστευση, απλοποίηση προκειμένου να μπορέσουν οι γεωργοί να χρησιμοποιήσουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προβλέπει η ΚΑΠΕ. Είναι Είμαστε βουλευτές, είμαστε οι άμεσα εκλεγμένοι λοιπόν από τους αγρότες και η απλούστευση γίνεται για τους αγρότες αυτούς ακριβώς. Και θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχουμε στη διαδικασία αυτή. Δεν μιλήσατε λοιπόν για τις γυναίκες γεωργούς. Έχετε στοιχεία, έχετε πληροφορίες. Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς ε, γίνεται, πώς είναι δυνατόν καμία χώρα έως τώρα να μην έχει καταρτήσει πρόγραμμα για τις γυναίκες αγρότες και τους νέους. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγιλέρα. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Το πρόβλημα της τάσης της Κομισιόν, της θέσης της Κομισιόν, είναι ότι χρησιμοποιεί κατάλληλο εργαλείο. Έχουμε πρόβλημα με τη διαδικασία. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι είναι μια διαδικασία που την χρησιμοποιεί ο Κατάινεν για να λύσει οικονομικά προβλήματα στο ΕΚΟΦΗΝ. Και η Κομισιόν για να επιλύσει άλλα προβλήματα. Χρησιμοποιώντας τα περιθώρια, οικονομικά περιθώρια που, και τα ποσά που περισσεύουν, ας πούμε, ε, από τη Γεωργία. Εμένα με ανησυχεί το θέμα της επικουρικότητας. Θα τη δώσετε για αυτή την πρόταση. Σε ό,τι αφορά τον ενεργό Γεωργό μπορεί να δημιουργηθούν τεράστιες ανισότητες. Μόνο αυτό ήθελα να πω, γιατί δεν έχω χρόνο, αλλά πάντως το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία εγκρίθηκε στο τέλος του χρόνου. Και είναι αστείο, είναι τόσο... Εμείς δεν πρόκειται να απεμπολίσουμε τα δικαιώματά μας. Έχουμε το δικαίωμα να εκφράσουμε γνώμη. Και αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι παράδεκτο. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Φυσικά, σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε με την ιδέα αυτή τη απλούστευση, αλλά στο έγγραφο που μας παρουσιάζεται ε, πρέπει να σας πω ότι έχω κάποιες αμφιβολίες. Αμφιβολίες τις οποίες θα ήθελα να αναφέρω σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ε, τα μεγαλύτερα επιδοτη, τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις προς τους νέους γεωργούς βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Κοιτάξτε, αυτό είναι αμφισβητήσιμο για παράδειγμα ως μέτρο στη χώρα μου όπου είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Το να υπάρχει λοιπόν μια υποχρέωση τέτοια είναι προβληματικό. Κάτι άλλο. Για την υποστηρίξη των μη γεωργικών παραγωγών που συνδέονται με τη γεωργία. Είναι όπνευτα γαλλικά. Τα οποία όμως ε, δεν έχουν ενδεχομένω ε, επιπτώσεις στο εισόδημα του Γιώργου και ως εκ τούτου ε, και αυτό είναι αμφισβητήσιμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 50% κατανομή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, τώρα, τώρα προτείνεται το 100% για την ευθύνη δηλαδή του κράτους μέλους. Αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο θεωρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπε. Είπατε απλούστευση. Αυτό μας προτείνετε; Προσυπογράφουμε αυτή την ιδέα. Όμως, να σκεφτείτε το εξής. Νομίζω ότι η καλύτερη απλούστευση είναι η σταθερότητα των κανόνων. Δεν πρέπει κάθε δύο χρόνια να αλλάζουμε τους κανόνες, όλοι θα συμφωνήσουμε αυτό. Αλλά αυτό συμβαίνει. Γιατί η γεωργία είναι μια μακροπρόθεσμη δραστηριότητα. Επομένω, τίθεται το εξή ερώτημα. Πρώτον, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, γιατί στη διαδικασία αυτή δεν εμπλέξατε περισσότερο το Κοινοβούλιο και επί της ουσίας. Όλα αυτά δεν είναι μία, ένας τρόπος για να, να αποσπάσετε την προσοχή μας από το βασικό, που είναι <laughs> η προετοιμασία της επόμενης ΚΑΠ και να αποσπάσετε την προσοχή και τη δική μας, αλλά και των γεωργών η κυρία Νταντσίλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, κύριε Επίτροπε, να σας ευχαριστήσω που ασχοληθήκατε με το θέμα της απλούστευσης της ΚΑΠ. Όπως διαπιστώσατε, σε όλες τις πολιτικές ομάδες έχουμε τον ίδιο στόχο. Ένα βασικός λόγος της περιπλοκότητας της ΚΑΠ είναι ότι έχουμε πολύ περίπλοκες βασικές πράξεις, βασικούς κανονισμούς δηλαδή. Σας ε, συγχαίρω λοιπόν για αυτή την προσπάθεια για απλούστευση. Όμως για να υπάρξει πραγματική απλούστευση της ΚΑΠ πρέπει να έχουμε σημαντικές πολιτικές αποφάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό η μέθοδος που θα επιλέξουμε. Όταν συνδυάζεται την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού με σημαντικές αλλαγές των τομεακών κανονισμών, δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη μέθοδος, δεν μπορούμε να τη δεχτούμε. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να υποφελέσει κάτι τέτοιο. Μία αναθεώρηση των τεσσάρων βασικών πράξεων στην ΚΑΠ θα πρέπει να γίνει φυσικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσά κύριε Επίτροπη, αλλά να εμπλέξετε και την Επιτροπή Γεωργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο φυσικά. Πρόκειται για νομοθετικέ πράξει που τι έχουν διαπραγματευτεί επί αυτά τα τρία θεσμικά όργανα με αυτή τη σύνθεση που σας είπα. Και ακόμη και αν η αθεώρηση έχει περιορισμένη εμβέλεια, θα πρέπει να γίνει με τους ίδιους φορείς, δηλαδή με τα ίδια όργανα που συμμετείχαν και στη διαπραγμάτευση του 2013. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι και η κατεξιότηση πράξης σε ό,τι αφορά τα μέτρα πρασινίσματος. Ελπίζουμε να τα λάβουμε αυτά τα μέτρα σύντομα για να τα εξετάσουμε και θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για αυτό το στοιχείο, για αυτό το στοιχείο το τελευταίο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Σύντομα. Κι εγώ είμαι αμήχανος μπροστά στην ε, διαδικασία που επιλέξατε. Φυσικά δεν συμφωνούμε όλοι, ή μάλλον συμφωνούμε όλοι, ότι πρέπει να απλουστεύσουμε. Και το είπατε κι εσείς πολλές φορές στις διάφορες ε, συναντήσεις μας, ότι πρέπει να γίνει η απλούστευση μεν, αλλά η απλούστευση θα αγγίξει λίγα πράγματα της ε, ΚΑΠ. Αλλά τώρα έχουμε τη διαδικασία Omnibus, που αφορά και τους τέσσερις βασικούς κανονισμούς της ε, ΚΑΠ και τους μεταρρυθμίζει. Συμφωνώ με την προλαλή σας. Υπάρχει το κείμενο και υπάρχει και το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι πολιτικό και δημοσιονομικό και νομίζω ότι αυτά που μας προτείνετε δεν νομίζω ότι είναι για τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ αυτή καθεαυτή, αλλά ε, αφορούν άλλα διακυβεύματα που ξεπερνούν την ΚΑΠ και τη γεωργία. Και στις δηλώσεις σας είπατε ε, θα πρέπει να μπουν όλα αυτά σε εφαρμογή το πρώτο, την πρώτη πρώτου του 18. Δηλαδή το 17 θα το περάσουμε όλοι, όλο να δουλεύουμε πάνω σε αυτή την ε, πρόταση που θα ακυρώσει δηλαδή και θα κρύψει τα ουσιαστικά προβλήματα που είχε η ΚΑΠ που πάει μέχρι το 20. Ακόμα και να απλουστεύσουμε, θα πρέπει να τα απλουστεύσουμε κατελάχιστον. Και δεν μπορούμε να κρύψουμε κάτω το χαλί τα βασικά διακυβεύματα τα οποία μας απασχολούν ε, σε ό,τι αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Ευχαριστώ, ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, συμφωνώ με το σχόλιο που υπόθηκε, να το ξαναπώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για ένα, να σταθώ σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Νομίζω ότι εκεί το παίξατε καλά, αλλά θέλω να ε, είμαι σίγουρος ότι το κατάλαβα καλά. Καταφέρατε να διατηρήσετε το σύνολο του προπολογισμού της ΚΑΠ, ε, ενσωματώντας και την ενίσχυση για τους μετανάστες στην ΚΑΠ. Σωστό. Το κατάλαβα καλά. Εάν ναι, είμαι ικανοποιημένο. Γιατί αποφεύγει ένα τμήμα του προπολογισμού τη ΚΑΠ να φύγει και να το χάσουμε διαπαντό. Όποιο και είναι ο αριθμό των προσφύγων που θα υποδεχθεί η Ευρώπη. Εάν ναι, Καλό θα ήταν να έχουμε αυτή την ενημέρωση, δεν την αναφέρατε καθόλου στην εισαγωγική σας παρατήρηση. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε ότι θα λειτουργήσουν τα πράγματα στην πράξη. Thank ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κέρδος και όχι τόσο πολύ η ρευστότητα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ένα από τους βασικούς στόχους είναι η προώθηση των οικονομικών ε, μέσων. Στο 2.02 λέτε να παραχθεί, ε, να δοθεί υποστήριξη μόνο σε όσους θεωρούνται ότι είναι βιώσιμοι. Δηλαδή, στην παρούσα φάση, αν είναι κανείς ε, εκτροφέας βοηου αν είναι κλεργητής δημητριακών ή γραφειοπαραγωγός, τι γίνεται. Το πρόβλημα είναι να αντιμετωπίσουμε φυσικά να αντιμετωπίσουμε τις αποτυχίες της αγοράς. Αλλά το έχουμε συζητήσει ιδιαίτερα το θέμα αυτό και έχουμε και μία συγχώνευση με, μεταξύ EBP και Slane και αυτό σημαίνει ότι 40% του τομέα των εγωπροβάτων θα αντιμετωπιστεί από το θέμα αυτό και 26,8% του τομέα του βοη κρέατος. Ενώ εκ παραλλήλου οι αγρότε επιτρέπεται να οργανώνονται μόνο σε επίπεδο 15%. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν τα προβλήματα στην Ιρλανδία. Αλλά ουσιαστικά είναι. Μιλάει με την η γλώσσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε και το άρθρο 207. Αναφέρεται ρητά την Ιρλανδία. Γιατί, τι σημαίνει θα μειωθεί τελικά η συνολική χρηματοδότηση της ε, Ιρλανδίας, ο κ. Ροπέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε, η ΚΑΠ θα πρέπει να εξασφαλίσει τη την επιβίωση των ε, αγροτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σας ευχαριστούμε, λοιπόν, Επιτρόπε, που θέλετε να απλοποιήσετε τους κανόνες για να υπάρξει ευελιξία. Αλλά οι φάκελοι ήδη έχουν κατανεμηθεί και δεν αρκούν, για παράδειγμα, για τις χώρες της Βαλτικής. Άρα η συνολική εικόνα μπορεί και να μην αλλάξει ιδιαίτερα. Σημειώθηκαν διάφορες κρίσεις. Στο γαλακτοκομικό κλάδο, στο χειρίο κρέας, τώρα σε ό,τι αφορά ε, τα δημητριακά, τα συντήρα. Είναι δύσκολο να επιβιώσουν οι αγρότες αυτοί. Ήλπιζα να σημειωθεί κάποια πρόοδο σε ό,τι αφορά την εναρμόνωση των πληρωμών για όλα τα κρατημέλη. Και θα ήθελα να το σχολιάσετε παρακαλώ αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γόιμπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Επιτροπέ. Αυτά που προτείνετε είναι μία κατάφορη παραβίαση των ε, μάλλον και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ε, Γεωργίας στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Και τι άλλο κάνετε με το Omnibus. Βάζετε την ε, βάση και αλλάζετε τη βάση για την επόμενη διαμόρφωση των επόμενων δημοσιονομικών προπτικών και για την επόμενη ΚΑΠ και μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Τώρα δηλαδή παρεμβαίνετε στην ανάπτυξη της υπαίθρου. Φεύγει από τα γεωργικά και πάει στα θέματα πολιτικής συνοχής αποδυναμώνεται την Επιτροπή μας. Μην σας πω ότι σκάβατε και τον ίδιο στο λάκκο, γιατί υπονομεύετε και τη δική σας ε, δύναμη Όταν η αναπτύξη του υπαίθρου, της αναπτύξης υπαίθρου διαχωριστεί από την αγροτική ανάπτυξη, αποδυναμώνουμε και την υπαίθρο, αλλά και τη γεωργία. Τι προγραμματίζετε λοιπόν να κάνετε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το ακούσω. Η ε, κυρία Νόχη. Σα ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ε, κύριε Επίτροπε, τι να σα πω, εγώ είμαι λίγο απογοητευμένη. Απογοητευμένη, πραγματικά απογοητευμένη. Δεν σα ε, εξέλεξα τότε, δεν σα ψήφισα τότε και ίσω καλά έκανα γιατί μα είχατε υποσχεθεί απλούστευσει, απλοποιήσει που δεν θα πλέξουν τη βάση και το περιεχόμενο, αλλά πραγματικές απλοποίησεις. Αυτά που έχουμε λοιπόν επιτάπητος για την ρύθμιση Omnibus, ε, δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω, καλά τα είπαν οι συνάδελφοι. Από την αμόντη επιτροπή μας. Αλλά για να επανέλθω σε κάποια άλλα ζητήματα περιεχομένου. Δεν μας δώσουν αυτές τις απλοποίησεις για τους κανόνες, για τα θέματα αυτά που μας απασχολούσαν, όχι θέματα περιεχομένου. Δύο χρόνια μας τα χρωστάτε αυτά. Και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη γιατί αυτό που καταφέρετε ως πρόταση είναι πρόταση αλλαγής της ουσίας της αγροτικής πολιτικής. Δεν έχουν να κάνουν αυτά με απλοποίηση. Μπαίνετε στο βασικό δίκαιο και στις τέσσερις βασικές νομοθετικές πράξεις παρεμβαίνετε. Άρα δεν εκπληρώνετε και την υπόσχεση που μας δώσατε ότι θα χρησιμοποιήσετε ό,τι περνάει το χέρι σας προκειμένου να υπάρξει απλοποίηση στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. 0% λοιπόν έχετε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις σας και τις δεσμεύσεις σας. Συμφωνώ και με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά αυτό σημαίνει παράλληλα ότι δεν έχετε προτείνει τίποτε για να προσταθεί το βασικό δικαίωμα. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Θέλω να ρωτήσω, δικιά σας η Γενική Διεύθυνση έχει προβεί σε κάποια έρευνα όσον αφορά ευάλωτους τομείς που μπορεί να χτυπηθούν από το Brexit, όλους ιδιαίτερος. Σίγουρα θα ξέρετε ότι ο πρώτος τομέας που απειλείται σοβαρά από ένα Brexit είναι στην Ιρλανδία η Γεωργία. Η μανιταροπαραγωγή ήδη από το 2013 υποφέρουν και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί θα βρεθούν σε ιδιαίτερο κίνδυνο. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο εσείς θα ζητήσετε από την γενική σας διεύθυνση να συνεργαστεί με τους Ιλλανδούς παραγωγούς έτσι ώστε να βοηθηθεί ο κλάδος ο οποίος δίνει και πολλή δουλειά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την δυνατότητα που μας δίνετε να συζητήσουμε σήμερα, γιατί ασκήθηκε πολύ κριτική για τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας παρακαλέσω ε, κάπως να μην υπερβάλλουμε κιόλα. Πρέπει σε κάποια φάση να γνωρίσουμε ότι στην μεταρρύθμιση της ΚΑΠ πολλά από αυτά που πρότεινε ο Επιτρόπος δεν λειτουργήσα και για να δώσω ένα Παράδειγμα, αποφασίσαμε να ορίσουμε τον ενεργό γεωργό. Αλλά αυτό στην πράξη σημαίνει, για παράδειγμα, ότι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται κοντά σε ένα κάμπινγκ δεν έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν επιδοτήσεις. Θα πρέπει όμως, και αυτέ οι επιχειρήσεις κάπως να επιβιώσουν. Νομίζω ότι ο σκοπό μας δεν είναι να δυσκολέψουμε τη ζωή των μικρών επιχειρήσεων, γιατί ακριβώς αυτές θέλουμε υποτίθεται να υποστηρίξουμε και να παραμείνουν σε μικρό επίπεδο, ε, όχι να τους βάλουμε κι άλλη μια α, κεραμίδα οικονομικά, δηλαδή να χάσουν τις επιδοτήσεις τους. Καλό θα ήταν λοιπόν να κοιτάξουμε λίγο και τις λεπτομέρειες και να σταματήσουμε τις ε, φλιαρίες, τις ιδεολογικέ ενδεχομένω και να κοιτάξουμε αυτά που προτείνονται προκειμένου όσα έχουμε αποφασίσει να περάσουν στην πράξη, να εφαρμοστούν και να μην παρατήσουμε στην τύχη τους, τους αγρότες μας. Αυτό θεωρώ ότι θα αποτελέσει το θέμα του μέλλοντος και γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι κύριε Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε συνδεθειμένος να έρθετε εδώ και νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε στο μέλλον καλύτερη εφαρμογή της ε, ΚΑΠ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμμερίζομαι πολλέ από τι παρατηρήσει που έκανε η προηγούμενη συνάδελφοι για τη διαδικασία Omnibus. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσφατη επίσκεψή σα στη Νότια Ιταλία, στη Σικελία και στην Καμπάνια. Είδατε από κοντά τα προβλήματα που έχει ο τομέα των προκυπευτικών τελευταία χρόνια. Ε, υπάρχει, χτυπάει το καπανάκι, υπάρχει απελπισία, απόλυτη απελπισία. Στη Σικελία ε, έχουμε έναν ιό που λέγεται Τριστέτσα, ο οποίος έχει γονατίσει τον κλάδο μα ανάγκασε ορισμένους ε, παραγωγούς να ξεριζώσουν ε, ε, λεμόνια, ελιές, πορτοκάλια κτλ. που αποτελούν σημαντικό τμήμα της οικονομίας του νησιού αλλά και εξασφαλίζουν και την διοπικιλότητα. Μα, ε, μας υποσχεθήκατε ότι θα εξετάσετε την κατάσταση. Τι θα πείτε, Επίτροπε, στου γεωργούς. Θα χρησιμοποιήσετε τις ρήτρε διασφάλισης. Ένα πακέτο βοήθειας προβλέπετε για την επίλυση αυτών των προβλημάτων στην Σικελία και στην Καμπανία. Δεδο, δεδομένως της, της ε, που υπάρχει. Τι, θα, τι να πούμε στους γεωργούς που επισκεφτήκατε. Ποια θα είναι η απάντηση της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ που είστε εδώ. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα άλλο για τα διαδικαστικά. Νομίζω ότι με κάλυψαν και σε Δύο θέματα θέλω να θίξω. Αυτά που αναφέρθηκαν σε ό,τι αφορά τις ασφάλειες είναι πολύ ενδιαφέροντα. Αλλά πολλά και σε έχω πει ότι υπάρχουν δυνατότητες απλούστευσης. Για παράδειγμα, στην ε, περιοχή μου έχουμε δεκάδες χιλιάδες ασφάλειες μικρών παραγωγών στα πλαίσια ενός ομίλου. Θα ήταν καλό λοιπόν να λαμβάνει ο ομίλος αυτός τα χρήματα αυτά. Αντί όμως να υπάρχουν 10.000 αιτήματα τα οποία να πληρώνονται, θα μπορούσε να υπάρχει πιο απλή διαμόρφωση του συστήματος. Και μία ερώτηση να σας κάνω. Προτείνεται σε κάποια κράτη-μέλη της Μέσης Ευρώπης, της Κεντρικής Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και το Λουξεμβούργο, ορίζεται 1% ενίσχυση από εθνικούς πόρους. Πώς ε, γίνεται αυτό. Μου φαίνεται λίγο περίεργο και αυτό δεν προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι λοιπόν έτσι εξαντλήσαμε το κατάλογο των ομιλητών, λέει ο Πρόεδρος. 30 άτομα πήραν το λόγο και νομίζω ότι θίξαμε όλα τα προβλήματα που είχαμε υπόψη μα. Κύριε Πέτραπε, να πάρετε το λόγο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό για εσάς. Όπως και να έχει. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά συνεπάγεται και μια τόσο σημαντική θέση όπως αυτή που κατέχετε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, πέρα. Εγώ δεν είμαι εδώ για να αποφασίσω ποια θα είναι η διαδικασία διαθεσμικά, το πώ θα αντιμετωπίσουμε τον μηχανισμό αυτό στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Η πρόταση αυτή έγινε από άλλου, όχι από εμένα, και εγώ απλά δράπαμε τη ευκαιρία για να προτείνω προτάσεις στα πλαίσια του Omnibus που θα μπορούσαν να περάσουν για να προωθηθεί η ατζέντα της απλούστευσης. Καταλαβαίνω και σέβομαι δε αυτά που είπαν όλοι για τη διαδικασία και είμαι διτεθειμένος να συνεργαστώ με την Επιτροπή ή όποια Επιτροπή αποφασιστεί ότι είναι η αρμόδια για να συμπληθεί η πρόοδος στις προτάσεις αυτές. Ε, συνεργάζομαι με την ε, Άγκρη και με μεγάλη μου χαρά. Αλλά αυτά τα αποφασίζουν άλλοι και υπάρχουν διαθεσμικές συζητήσεις οι οποίες ε, κατέληξαν στις αποφάσεις αυτές. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τα αποφασίζουν αυτά, αλλά εγώ είμαι διτεθειμένος να εργαστώ στα πλαίσια του όποιου μηχανισμού έχω στη διάθεσή μου. Νομίζω ότι οι προτάσεις που έχουμε εδώ ανταποκρίνονται σε κάποιες από τις επιθυμίες σας. Δεν λέω ότι είναι το τελειωτικό βήμα αυτό, το οριστικό, το ιδιωτικό πακέτο και τελείωσε μετά. Νομίζω ότι οι διάφοροι συντονιστέ το ανέφεραν αυτό και το σέβομαι. Και τα μεταφέρω τα μηνύματα αυτά προ την Επίτροπο για Θέματα Προπολογισμού. Ο κ. Ρίγο αναφέρθηκε στη δυνατότητα βελτίωση των εμπορικών σχέσεων και με τη Ρωσία. Εγώ με μεγάλη μου χαρά να επανέλθω σε φυσιολογικά επίπεδα οι εμπορικές σχέσεις με την ε, Ρωσία συναντήθηκα και με εκπροσώπου. Αλλά αυτό είναι θέμα του Συμβουλίου Εκτορικών Υποθέσεων. Αν θα άρουν ή όχι τις κυρώσεις. Αυτή είναι άλλη συζήτηση. Ε, μέχρι να γίνει αυτή η οχι τι κυρωσει πώς εγώ να κάνω το οτιδήποτε. Ο κύριος Χόσλινγκ. Δεν υπάρχουν χρήματα για... για μαθήματα γκολφ. Και αν κάποιο παίρνει χρήματα για δραστηριότητε που δεν είναι αγροτικέ, πολύ απλά παραβιάζει του νόμου. Δεν ξέρω τι λέτε εσεί, αλλά είναι λάθο πολύ απλά αυτό. Έχουμε πιο εύκολα συστήματα μεταβολή και τοποποίηση του προγράμματο ε, ανάπτυξη τη υπέτρου για τη συμμετοχή κάποιων τομέων με το εργαλείο σταθεροποίηση εισοδημάτων. Αυτά λοιπόν μπορεί να επιτευχθούν αρκετά γρήγορα σε κάποιες περιφερειές από τις τοπικές κυβερνήσεις αν επιθυμούν πραγματικά να τροποποιήσουν τα εργαλεία αυτά μπορούν μέσα σε δύο-τρεις μήνες να το κάνουν αυτό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Και η δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων αυτών είναι επίσης κάτι αρκετά εύκολο αν λάβουμε έγκριση. Φυσικά όλα τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν μέσω του συνομοθέτη να απορριφθούν αυτές τις προτάσεις ή να προσθεθούν. Να σας ε, υπενθυμίσω ότι εσείς κάνετε εκστρατεία να βγείτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις επιπτώσεις τώρα. Είναι δύσκολες οι επιπτώσεις και καταλαβαίνω ότι δυσκολεύεστε στον Ευρωπαϊκό Βασίλειο. Ακόμα διάφορες απόψεις από διάφορους υπουργούς, από διάφορους ε, ηθήνοντες για το ποιε θα είναι οι συνέπειες. Θα δούμε, θα δούμε στο επόμενο διάστημα και θα γίνουν διαπραγματεύσεις αλλά πολλά θέματα θα έχουν να κάνουν και με τη γεωργία και ελπίζω Πρόσφατα προτάθηκε να υπάρχει μεταφορά χρημάτων από τον τομέα της γεωργίας στον τομέα της υγείας. Ελπίζω να μην περάσει αυτό για τους γεωργούς σας, γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι δυνάμεις θα κινητοποιήσετε για να μην συμβεί αυτό. 95% της ε, γης ε, των αεροτρέων γεών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποιο σκοπό θέλει ο αγρότης, αν θέλει κανείς να παράγει πρωτεϊνούχα. Για παράδειγμα, μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά έχουμε και στόχο 5% για οικολογική καλλιέργεια και έκανα μία πρόταση προκειμένου η πολιτική αυτή της ΚΑΠ να τονιστεί όχι μόνο η οικονομική της διάσταση, αλλά και η περιβαλλοντική της διάσταση, η κοινωνική της διάσταση, για να υπάρξει και προστασία της βιοπικιλότητας. Με τον τρόπο τον οποίο αποσκοπούσαν και οι αρχικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατέθεσα λοιπόν μια τέτοια πρόταση, την τροποποιώ την πρόταση από την αρχική, αλλά κρατώ την, ε, το βασικό στόχο σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τη χρήση λιπασμάτων, ζυζανεκτών κτλ. Και μου κάνει εντύπωση ότι και η κυρία η οποία υποστήριξε αρχικά αυτή την πρόταση τώρα έρχεται και κάνει το σχολείο που έκανε. Δεν υπάρχει δισταγμός για το φίλο εκεί να χρησιμοποιηθούν ε, δάνεια για να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις. Έχουμε ήδη την ελαστικότητα και την ομοθεσία για να γίνει αυτό και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές χώρες μέλη και η Ιρλανδία που έχει κάνει προτάσεις για μόχλευση της αρρωγής που υπογράμμισα για όλες τις χώρες ε, μέλη ήδη τον Ιούλιο. Αλλά για να γίνει αυτή η μόχλευση θα είναι 2,9%. Hm? Το επιτόκιο. Αν θέλετε να διπλασιαστεί, αν το Υπουργείο θέλει να το κάνει, μπορεί. Νομίζω ότι είναι πράγματι καλό να μπορούν να πάρουν παραπάνω χρήματα οι γεωργοί και τα μέτρα αυτά να ληφθούν υπόψη σε αυτά τα πλαίσια. Τώρα το 267. Είναι υπέρ της Ιρλανδίας κύριε Φλάνναγκαν, γιατί είναι 100% σε χρηματοδότηση μια που ήταν σε πρόγραμμα Ιρλανδία. Τέλειωνε το 2016, ενώ το Omnibus, με το Omnibus θα τελειώσει στο τέλος της ε, περίοδου πολιτών δημοσιονομικών προπτικών. Κύριε Κάρτιρ, ξέρω τα προβλήματα που έχει η Ιρλανδική ε, Γεωργία. Ήμουν σε αντιπροσωπή του κόμματό σα χθε, όπω ξέρετε, και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Και δουλεύουμε παρασκηνιακά σκληρά για να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε διαπραγματεύσεις λάβουν ε, χώρα στα πλαίσια του Brexit. Σίγουρα και η γεωργία θα συμπεριληφθεί, όπως και οι εμπορικές σχέσεις. Μπορεί να είναι δύσκολα για την ε, Ιρλανδία και την Βόρεια Ιρλανδία, όπου υπάρχει εκατομμύρια γάλακτος που καθημερινά περνάνε από την Βόρεια στην Νότια Ιρλανδία. Η πίεση είναι τεράστια. Αν ένα τομέα σχέται σε δυσκολία, μια χώρα μέλος μπορεί να σκεφτεί και να εισαγάγει προσωρινά μέτρα με εγγυήσει, με δάνεια από την κυβέρνηση. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και η Ιρλανδία λοιπόν μπορεί να το κάνει με το επίπεδο αντεμίνιμους. Ο ενεργός αγρότης, πολλοί αναφέρθηκαν σε αυτή την έννοια. Η πρόταση της Επιτροπής είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που εσείς αποφασίζετε ως ε, συνομοθέτες. Και ήταν ε, δύσκολο έτσι κι να το λύσουν οι συνομοθέτε. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα αρνητικό κατάλογο. Εγώ προσπαθώ να λύσω το πρόβλημα που έχει προκύψει μέχρι σήμερα, δίνοντα περισσότερη ευελιξία στι χώρε μέλη να αποφασίζουν από μόνες του. Μπορούν να δεχτούν τον ορισμό, να τον αρνηθούν τον ορισμό, να τον τροποποιήσουν τον ορισμό του ενεργού αγρότη. Ήταν μεγάλη δυσκολία για πολλές χώρες μέλη ορισμό αυτός και σε αυτό προσπαθήσαμε εμείς να βοηθήσουμε. Τώρα για τον προπολογισμό και τα όρια. Κύριε Νταντά, κυρία Ράντς Γκαρσία, 20-20 είναι τα όρια και δεν τίθεται θέμα αλλαγής. Τα χρήματα είναι όσα ήταν. Το 2% το όριο που είναι για τους νέους αγρότες είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο βάσει της νομοθεσίας. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραμανώ, αλλά το 2% του προπολογισμού θέλω να φροντίσω όντω να πηγαίνει σε αυτούς. Υπήρξαν προβλήματα σε κάποιες χώρες μέλη. Ο κύριος Μπούντα αναφέρθηκε στις οργανώσεις των παραγωγών. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με κάθε δυνατό τρόπο συζητήσεις μαζί τους με τις οργανώσεις των παραγωγών και θα το δείτε αυτό όλο και περισσότερο όταν αρχίσουμε να συζητάμε τον Ιανουάριο με τη Task Force εδώ στην Επιτροπή σας για καλύτερες ε, διαπραγματεύσεις και θα στηρίξουμε τις οργανώσεις των παραγωγών στις χώρες. 14% σε μια χώρα ε, συμμετέχουν στις συλλογικές συμβάσεις. Χρειάζονται περισσότερα. Ο κύριος Έρντος αναφέρθηκε επίσης στον προπολογισμό. Σας είπα, ε, έχει καθοριστεί 2020, αλλά κοιτάμε μήπως μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο για τις αρδρευόμενες επιφάνειες. Συνεργαζόμαστε με τον κύριο Βέλε την GE Περιβάλλοντος για να βοηθήσουμε τον τομέα των τροφίμων και άλλους κλάδους που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης και χρειάζονται πολύ νερό. τον Ιανουάριο του 2017 θα έχουμε κάποια έκθεση μεταξύ μας για αυτά τα ζητήματα. Πολλοί αναφέρθηκαν στην απογοήτευσή τους από την εφαρμογή. Μα ναι, και γι' αυτό προσπάθησα τα τελευταία δύο χρόνια να τα διορθώσω. Και στην κυρία Μάκαλς και στον Μητεπίνης. 270 μέτρα έχουν, 270 μέτρα έχουν ε, εφαρμοστεί και τώρα αρχίζουμε να κοιτάμε πώς προχωράνε αυτά. Δεν δέχομαι ότι εγώ δεν τήρησα τις υποσχέσεις μου. 270 μέτρα και θα κάνω και περισσότερα μετά τη μεταρρύθμιση 2020. Θα προτείνουμε στη δημόσια διαβούλευση διάφορες προτάσεις για να δούμε τι θα κάνουμε στον επόμενο γύρο εφαρμογή της ΚΑΠ μετά από το 2020. Θα αρχίσει αυτή η διαδικασία λοιπόν σύντομα και φυσικά και θα συμμετέχετε κι εσείς. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας από την εφαρμογή γιατί έτσι καλλιώς πρόκειται για συμβιβασμό. Οι προτάσεις είναι συμβιβασμό. Ξέρετε ότι χιλιάδες τροπολογίες είχαν υποβληθεί. Φυσικά και υπάρχει η διάσταση απόψεων επειδή είναι περίπλοκο το θέμα. Θα συνεχίσουμε όμως να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας για να λύνονται αυτά τα προβλήματα με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο. Η κυρία Γκίλη επίσης αναφέρθηκε στο λάθος εργαλείο. Δεν ξέρω, εγώ προσπαθώ να χρησιμοποιήσω το εργαλείο το οποίο μου προτάθηκε και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με αυτό για να υπάρξει απλοποίηση. Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα. Εγώ θέλω να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Αλλά αν θέλετε κάτι άλλο, εσείς θα το δείτε αναφέρθηκε και η ρύθμιση του 50-50. Γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι προκειμένου να κτηθούν χρήματα από χώρες μέλη για να προστατεύσουμε τον κοινοτικό προπολογισμό. Υπάρχει η διαδικασία που το δεύτερο 50% παίρνει χρόνια για να ανακτηθεί. Η διαδικασία κρατάει πάρα πολύ και πρόκειται για χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Καλύτερα λοιπόν να είμαστε στο 100% παρά να περιμένουμε για χρόνια να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ανακτηθούν τα χρήματα. Για το greening, το πρασίνισμα, πρότεινα 15 διαφορετικές προτάσεις της ομάδας εμπεριγνωμόνων. Διευκρίνηση διαφόρων ζητημάτων που δυσκολεύουν τους αγρότες. Αλλά περιλαμβάνεται και η, και εφαρμογή της απαγόρευσης των παρασιτοκτόνων σε ε, ορισμένες ως οικολογικές περιοχές. Χρειάζεται και άλλη δουλειά στις ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα συνεχιστεί αυτό το μήνα. Αλλά καταλήγεται σε συμπεράσματα χωρίς να πρέπει τη Δευτέρα το Συμβούλιο λέτε ε, ήθελε να απορρίψει την πρότασή μου. Μα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Δέχονται να παραμείνει η απαγόρευση αυτή. Κύριε Φλάνεγκαν, για την αποτυχία της αγοράς 1,5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν από τα χρήματα των φορολογούμενων και άλλα 56 δις για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν ήταν εύκολο, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με τα οικονομικά μέσα είναι μόχλευση των χρημάτων αυτών. Άρα με δάνεια να βοηθήσουμε με καλούς όρους, όπως στην Ιρλανδία, και 2.000 άνθρωποι εξέφρασαν ενδιαφέρον. Υπάρχει επιλογή. Δεν είναι υποχρεωτικό φυσικά. Αν μπορείς να πάρεις με 3 με 4% φυσικά είναι προτιμότερο από το 6-7%. Οπότε πρέπει να βρούμε νέους μηχανισμούς για να βρούμε χρήματα και να βοηθήσουμε τους αγρότες που θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Όσοι θέλουν να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις, δηλαδή πρέπει να μπορούν. Είναι δύσκολο για τους συνεταιρισμού να έχουν χρέος όταν οι τράπεζες δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Το μέσο σταθεροποίησης είναι ένας άλλος τρόπος, πέρα από τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Οι υπουργοί, το πανεχτές και ο υπουργό στην Ολλανδία, είπε για τα 150 εκατομμύρια για να βοηθηθεί ο τομέας. Αυτές είναι επιλογές λοιπόν που υπάρχουν για τους υπουργούς και μπορούν να τις εφαρμόσουν. Ο κύριος Τεντέν ρώτησε για τη μετανάστευση, για την ασωμάτωση της ΚΑΠ στο μεταναστευτικό. Είπαμε ότι γι' αυτό γίνονται αλλαγές μεταξύ άλλων. Υπάρχουν λόγοι στις ε, αγροτικές περιοχές που στηρίζουν γιατί ε, μπορούν να βοηθηθούν. Πρόεδρε, για το προκυπευτικά. Με ρωτήσατε. 395 εκατομμύρια δαπανώνται προκειμένου να βοηθήσουμε τον κόσμο στα οποροκυπευτικά για να αντιμετωπίσει το εμπάργο, το ρωσικό έγινε επέκταση και για τον επόμενο χρόνο. Αλλά αυξήσαμε και την απόσυρση. Πολλοί το ρώτησαν, οι Ισπανοί, οι Ισπανικοί συνεταιρισμοί και είπαμε ότι θα συνεχίσουμε και το 2018. Νομίζω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να δώσουμε κάποιο αντιστάθμισμα. Δεν μπορεί να μην είναι αρκετό, αλλά πρέπει να αναγνωριστεί ότι χτυπήθηκε πολύ αυτός ο κλάδος. Βέβαια, πρέπει να βρεθούν και νέες ευκαιρίες. 32 χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στοχεύτηκαν προκειμένου να έχουμε πρόσβαση και σε αυτές τις αγορές. Αυτό χρειάζεται. 32 λοιπόν είναι μεγάλη επιτυχία. Ολοκληρώνω με το εξή. Ο ρόλος της ε, πολιτικής της υπαίθρου, ξέρω ότι το έχετε διαβάσει, 355 ενδιαφερόμενοι ήρθαν στη διάσκεψη και έτσι πιστεύω μπορούμε να βοηθήσουμε για τη βελτίωση τη ζωή στην Ήπεθρο. Θα το κάνουμε και στο μέλλον. Ελπίζω ότι βγαίνουν λογικά συμπεράσματα και από τη διάσκεψη αυτή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συγγνώμη, Επίτροπε, για την παρέμβασή σας. Ο κύριος Ντάσος θέλει ακόμα να κάνει μια ερώτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Διαπιστώνω. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία, εμείς στο Κοινοβούλιο μπορούμε να αποφασίσουμε μαζί με το Συμβούλιο από κοινού. Και κύριε Επιτροπέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι ε, επιλέξατε μια ρύθμιση η οποία μας επιτρέπει να τράσουμε γρήγορα. Όλα τα υπόλοιπα επαφίονται σε εμάς, εκτρώνται από εμάς. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Επιτροπέ. Ε, δεν απάντησα μια ερώτηση που έγινε για τις ασφάλειες. Ε, εξετάζουμε όλα αυτά τα θέματα στα πλαίσια της ε, Task Force ε, και της έχεις προετοιμάσει για τις uh, γεωργικές αγορές. Θα δούμε ποια είναι τα επιπλέον εργαλεία που χρειαζόμαστε, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε αθεκτικότητα ε, στις γεωργικές αγορές. Είναι σημαντικό αυτό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους γεωργούς, ορισμένε από τις προτάσεις χρειάζονται, ε, από αυτές τις προτάσεις χρειάζονται τροποποίησεις. Εάν υπάρχει κάτι στις ε, πρακτικές των ξένων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, κανένα πρόβλημα να πάρουμε τις λεπτομέρειες και να προσαρμόσουμε αυτές τις προτάσεις στη δική μας πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Το πιο σημαντικό είναι η δημοσιονομική σταθερότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση σε πολλοί αριθμέ αγορές και στο γαλακτοκομικό τομέα, στο χείριο κρέας, στα οποροκυπευτικά, στα σιτηρά και φυσικά γνωρίζουμε και τις διάφορες δράσεις που ε, προωθήθηκαν το περασμένο φθινόπωρο και φέτος το καλοκαίρι. ήψους ε, ύψους ενός εκατομμυρίου και πλέον ευρώ με σκοπό να ενισχυθούν και να στηριχθούν οι γεωργοί. Σε ό,τι αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων για την πρόταση Omnibus. Υπάρχει η θέση του Κοινοβουλίου από τη μία, δηλαδή η θέση της Επιτροπής Γεωργίας για το πολιτικό σκέλος. Η Επιτροπή Γεωργίας ως αρμόδια για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα ήθελε να συνεχίσει να είναι ένας από τους βασικούς φορείς που θα συζητήσουν αυτό το θέμα. Βλέπω ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών θέλει το λόγο. Σας δίνω το λόγο, πρόεδρε. Κύριε πρόεδρε, ε, παίρνω το λόγο ως μέλος της Επιτροπής ε, Γεωργίας που προδρεύεται. Απλώς είμαι και πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όλα τα σχόλια που άκουσα, όλες τις ανησυχίες που εκφράστηκαν Και να σας πω τι θα πω στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Ε, εμείς λάβαμε από την Κομισιόν ένα κείμενο το οποίο ε, εκπονήθηκε λόγω του ότι ε, γίνεται μια ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτή ήταν και η δέσμευση που είχαμε λάβει το φθινόπωρο το 2013, ούτως ώστε να μπορέσει το Κοινοβούλιο να συμφωνήσει με το δημοσιονομικό πλαίσιο είχαμε πει ότι δεν θα το δεχόμαστε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μόνο εφόσον μπορούσαμε το αναθεωρήσουμε στα μέσα της διαδρομής. Εδώ είμαστε, στα μέσα της διαδρομής. Και η Κομισιόν θέλησε να προσθέσει μια σειρά από μηχανισμούς, μια σειρά από εργαλεία, με σκοπό την απλούστευση. Και όλα αυτά τα συμπεριέλαβε σε ένα κείμενο που το λέει Omnibus. Λοιπόν, τι διαδικασία θα ακολουθήσουμε τώρα στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, που είναι αντικείμενο τη αναθεώρηση που θα την εξετάσουμε μαζί με το σχέδιο προπολογισμού του 2017, ούτω ώστε να υπάρχει μια καλή έτσι, συνάφεια ανάμεσα στον προπολογισμό του 2017 και στην αναθεώρηση του πολιετού δημοσιονομικού πλησίου και να λάβουμε υπόψη τον διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμό 4 του 2016, που στην πραγματικότητα αναδιανέμει 8 δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη-μέλη. Και φαντάστε την ανυπομονησία των κρατών μελών να πάρουν το μερτικό τους από αυτά τα 8 δις. Επομένως, θέλουμε αυτά τα τρία κείμενα να τα δούμε σαν πακέτο. Σε ό,τι αφορά το Omnibus, που ήταν το αντικείμενο των σημερινών σχολείων μας και που το σχολίασε και ο Επίτροπος, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιανουαρίου του 2017, ούτω ώστε το κείμενο να μπορέσει να εφαρμοστεί τελικά 1η-1η-18. Έχουμε χρόνο λοιπόν. Επί της ουσίας, ο στόχος είναι να φτιάξουμε μια κοινή επιτροπή, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, η Επιτροπή επίσης Προπολογισμών, με βάση το άρθρο 55 του κανονισμού. Και φυσικά να εμπλέξουμε και, την ε, Ευρωπαϊκή, και τις ε, επιτροπές που επηρεάζονται από κάποιες από τις διατάξεις αυτής της τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού και από τις τομεακές, ε, τα τομεακά θέματα. Πέντε εξειδικευμένες επιτροπές εμπλέκονται πέρα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών και Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Το να εμπλέξουμε όλες αυτές τις επιτροπές με βάση το άρθρο 55 στα πλαίσια μιας μεικτής επιτροπής σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεδριάζουμε ουσιαστικά στην αίθουσα της Ολομέλειας. Και καταλαβαίνετε ότι θα είναι πολύ απλό αυτό. Η πρόταση λοιπόν που είναι επιτάπητο σήμερα είναι να εμπλέξουμε όλες τις εξειδικευμένες επιτροπές και την Επιτροπή Γεωργίας με βάση το άρθρο 54 με μία αποκλειστική αρμοδιότητα για όλες τις διατάξεις που αφορούν όλος ιδιαίτερο την Επιτροπή ε, Γεωργίας. Τώρα, το θέμα που τίθεται είναι τι γίνεται στον τριμερή διάλογο, τι θα γίνει. Νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου ο εισηγητής της εξειδικευμένης επιτροπής θα, συνδεθ, θα εμπλακεί στη συζήτηση. Θα, δηλαδή θα έχουμε την Κομισιόν, το Συμβούλιο και τον συγκεκριμένο εισηγητή της κάθε επιτροπής. Θέλουμε να δούμε αν όλα τα κείμενα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο, το οποίο είναι βαρύ, έτσι. Είναι 280 άρθρα σε 300 περίπου σελίδες. Δεν είναι δηλαδή κάτι απλό που το ξεπετάμε έτσι. Υπάρχουν δύο ε, μέρη. Μία απλή αναθεώρηση της, του δημοσιονομικού κανονισμού και ένα δεύτερο τμήμα που αφορά τις διατάξεις τις τομεακές, έτσι. Τι πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι το σύνολο αυτών των διατάξεων να συνεισφέρει στην απλούστευση. Αν έχουμε διατάξεις άλλου τύπου, ίσως η Κομισιόν θα μπορούσε τη σοφία της να φανταστεί ένα άλλο μέσο, ούτως ώστε να επιτρέπει στις εξειδικευμένες επιτροπές να μπορούν να τα σκεφτούν αυτά τα πράγματα πριν αποφανθούν. Εκεί φτάσαμε. Ελπίζω ότι αυτά τα λόγια θα διασκεδάσουν κάποιες ανησυχίες που εκφράστηκαν. Η συζήτηση έχει ανοίξει και φυσικά η Επιτροπή Προπολογισμών είναι πολύ προσεκτική και λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Εν μέρη εξηγεί, εν μέρη καθησυχάζει. Η διαδικασία που προτείνεται ποτέ δεν είχε προχωρήσει σε τέτοια κλίμακα. Βέβαια πάντα υπάρχει μια πρώτη φορά για τα πάντα. Ελπίζουμε στη συζήτηση αυτή θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια διατύπωση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά για όλα αυτά τα τόσο σημαντικά ζητήματα για την Επιτροπή Γεωργίας. Ο κύριος Δεκάστρο. Θέλω και εγώ να υποφεληθώ από την ε, ευγένεια του προηγούμενου ομιλητή για να πω δύο λόγια. Μετά από αυτά που είπε, τον ευχαριστώ για αυτά βέβαια, και για την, ε, τον ευχαριστώ και για την ακρίβειά του. Δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο και λιγότερο επικίνδυνο χρονικός πώς να βάλουμε τα γεωργικά θέματα σε αυτόνομο κανονισμό. Είναι θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον προπολογισμό. Όπω ακούσατε από τη συζήτηση, Πρόεδρε, εδώ μιλάμε για ενεργό γεωργό, μιλάμε για νέους γεωργού. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον προπολογισμό, είναι συγκεκριμένοι κανόνες. Εάν καταφέρουμε να τα χωρίσουμε αυτά, τότε θα είμαστε και πιο γρήγοροι ω Κοινοβούλιο και θα σεβαστούμε το σφιχτό χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ωραία. Όλα συζητιούνται. Είναι βέβαια σαφές ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Δεν θα πάμε την πρωτοβουλία αυτή ως Επιτροπή. Θα προετοιμάσουμε όμως έγγραφα ώστε να ενημερωθούν όλοι στο Κοινοβούλιο. Μα επίσημα ε, μέσα Νοεμβρίου θα μας ε, ζητηθεί συνέχεια. Οπότε εμείς προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά ώστε να μπορέσουμε να εργαστούμε κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και να πετύχουμε τους επιθυμητούς στόχους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ακούγεται καλά. Ελπίζω οι προσκεκλημένοι μας στη σημερινή συνεδρίαση να το άκουσαν ακόμα καλύτερα. Θα είδαν στη συνεδρίασή μας πώς σκεφτόμαστε και πώς συζητάμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση λοιπόν, ευχαριστώ και τον Επίτροπο και όλους τους παρόντες. Αύριο μην ξεχάσετε να φέρετε τις κάρτες σας για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία στις 9 αύριο το πρωί. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε και τον Επίτροπο και όλους τους συμμετέχοντες.